Σας παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εκ μέρους όλων των μελών ε, της Επιτροπής Ήτρα για αυτή την ακρόαση για την οριζόντα 2020. Θα ήθελα καταρχήν ε, να καλωσορίσω όλους όσους ε, ήρθαν ε, από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης και από τις Ηνωμένε Πολιτείες, η συνεισφορά τους, χάρη και για τη συνεισφορά τους χάρη στη μόρφωσή τους στον ακαδημαϊκό τομέα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και τους προσώπους των κρατών μελών του Συμβουλίου, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλους τους θεσμούς που συμμετέχουν στη συζήτηση για τον ορίζοντα 2020 ε, την, ε, επίτρο, την αρμόδια επίτροπο, την ε, κυρία Κουίν και τον εκπρόσωπο για την Προεδρία της Δανίας, τον μόνιμο και μάλλον ο εκπρόσωπος της Προεδρίας της Δανίας και ο μόνιμος γραμματέας ε, θα έλθουν στη συνέχεια. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τους διάφορους εκπροσώπους ε, των πανεπιστημίων, των οργανώσεων για την έρευνα και του βιομηχανικού τομέα που έχουν έλθει από όλη την Ευρώπη και Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω ένθερμα τους εκπροσώπους του τύπου. Δεν ε, είναι έκπληξη που τόσα άτομα απάντησαν ε, στην πρόσκλησή μας ε, και προσέτρεξαν στις Βρυξέλλες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. οριζόντα 2020 είναι το τρίτο πιο σημαντικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από τα προγράμματα για τη Γεωργία και για τα διαφορετικά ταμεία σε ό,τι αφορά του χρηματοοικονομικού πόρου με ε, κονδύλια περίπου 80 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα θα καταστεί το πλέον σημαντικό για την έρευνα στον κόσμο. Αλλά το πιο σημαντικό ε, είναι ότι ο ορίζοντας 2020 είναι ότι πρέπει να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα για το μέλλον. Ε, οι πόροι ε, που θα εκταμιευθούν αποτελούν μια μεγάλη επένδυση ε, στο πιο σημαντική για της Ευρώπης, όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και όλο το Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι οι επιστήμονες μας είναι πιο σημαντική πηγή, ο πιο σημαντικός πόρος για την Ευρώπη. Εμείς ε, ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος ε, ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο για αυτούς ε, τους εγκεφάλους. Ε, εμένα με εξέπληξαν τα σημαντικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Μία πρώτη αξιολόγηση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μας έδειξε ότι και άλλα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ερευνάς αποκαλύφθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αλλά ταυτόχρονα έδειξε και ποια είναι τα δύναμα σημεία που δεν μπορούμε να δεκτούμε, το χάρη σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε εξαιρετική σε όλους τους τομείς της έρευνας και της ενέργειας και όπου χρειάζεται και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο ε, όπως και στη βιομηχανική τεχνολογία πρέπει να είμαστε επιτυχείς σε όλο το μέτωπο της καινοτομίας. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα πλαίσιο, για το ειδικό πρόγραμμα για το ορίζοντας 2020, καθώς και για τους κανόνες ε, συμμετοχής, ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας ε, και Έρευνα και για το πρόγραμμα Ευρατόμ. Δεν υπάρχουν αμφιβολίε ότι πρόκειται για ένα πολύ ευρύ πρόγραμμα, αλλά είμαι πεισμένη ότι θα αξίζει τον κόπο. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας ε, στον κοινοβουλευτική διαδικασία. Τα κύρια τμήματα του ΙΣΔΕΣΜΙΣ ορίζοντα 2020 υπόκειται σε μια διαδικασία συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα διαπραγματευτούν το πρόγραμμα και στο τέλος θα λάβουν μια απόφαση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε πολύ προσεκτικά αυτή την ε, πολύ σημαντική συζήτηση εμείς λάβαμε την έκθεση της συναδελφού της κυρίας Κερβαλίου, για την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης, την έκθεση του κυρίου Δ για την ε, προσωρινή αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου και την έκθεση της κυρίας ε, Ματίας ε, για την πράσινη χαρτά για το νέο πρόγραμμα που ονομάζεται τώρα Οριζόντες 2020 σήμερα. θα συζητήσουμε βάση μιας έκθεσης της Επιτροπής και θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εσωτερική συζήτηση με την Επιτροπή Ήτρε το φθινόπορο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που μάλλον θα ολοκληρωθούν ε, το πρώτο μίση του 2013 ή ακριβώς πριν ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα στις αρχές του 2014 μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με την έρευνα η Επιτροπή Ήτρε και η Ολομέλεια δήλωσαν πέρσι ότι η αύξηση του προπολογισμού για την έρευνα και την κοινοτομία μπορούν να ε, συνεισφέρουν στην αηφόρο ανάπτυξη αυτό σημαίνει ότι εδώ είστε μεταξύ φίλων δεν χρειάζεται να πείσετε την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ότι η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία είναι αποφασιστικέ για το μέλλον μα. Το γνωρίζουμε. Ζητούμε μόνο τη συνεισφορά σα για να προσδιορίσουμε τι προτεραιότητε και τις του καλύτερου όρου για το πρόγραμμα πλαίσιο. Θέλουμε ορίζοντα 2020 να ε, είναι ιδιαίτερα επιτυχή στην ιστορία της Ευρώπης και να ανοίξει τις πόρτες για το μέλλον της Ευρώπης. Η σημερινή ακρόαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού τέτοιες ε, σκέψεις με οδηγούν στο τελευταίο σημείο. Να αναφερθώ στο οργανωτικά. Η σημερινή ακρόαση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε μια μεγάλη αίθουσα, αλλά ίσως ε, να μην μα χωράει όλου. Έτσι λοιπόν, έχουμε και μια αίθουσα ακρόαση στην 1Ε2, όπου μέσω του διαδικτύου μπορεί κάποιο να ακούσει την ακρόαση και όλες οι παρουσιάσεις ε, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ιστοσελίδα της Επιτροπής Ήτρε μετά την ακρόαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας, ε, ε, αγαπητοί ομιλητές, αλλά πρέπει να υπάρχει και λίγος χρόνος ε, για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Βουλίου. Εγώ θα προσπαθήσω να γίνει σεβαστός ο χρόνος, έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στα 10 λεπτά και τα μέλη του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομοι στη χρήση του χρόνου στις ερωτήσεις, γιατί θα έχουμε 25 λεπτά για τις ερωταπαντήσεις κατόπιν κάθε πάνελ και θα δώσω δύο, λεπτό, δύο λεπτά σε καθένα για ε, τις ερωτήσεις ε, και σας παρακαλώ ε, θα ήθελα να ομαδοποιηθούν όλες οι ερωτήσεις ε, και να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές ε, για την απάντηση. Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Και τώρα θα δώσω το λόγο για το πρώτο πάνελ ε, σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες στην ε, κυρία Αριέρα Μαδουρέλ, ε, η οποία είναι η συγγήτρια για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κατόπιν αυτής της σημαντικής η εισήγηση που κάνετε, Πρόεδρε, όσον αφορά το σύνολο του προγράμματο Ορίζοντα 2020, εντάχει να σα κάνω και εγώ την ε, ε, εισήγησή μου για το πρώτο πάνελ και πρόκειται να δουλέψουμε σήμερα το πρωί έντονα. Και σε αυτό το πρώτο πάνελ πρόκειται να συζητήσουμε την πρώτη από τις τρεις προτεραιότητες αυτού του προγράμματος. Πρόκειται για αυτό το οποίο ονομάζεται άριστη επιστήμη. Μιλούμε όμω για την αριστεία της έρευνας και των ερευνητών μας. Επίσης θα συζητηθεί το τι θα κάνουμε ούτω ώστε να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια για να είναι επομένω η παγκόσμια κλίμακα πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Η αριστεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τι συζητήσεις για την έρευνα και τις επιστήμες. Πρόκειται για μια έννοια η οποία θεωρείται συνώνυμο της ε, πάρα πολύ καλής ε, ποιότητας κάτι δηλαδή το οποίο για ορισμένους είναι αμφίσιμο, δεν είναι τόσο σαφές και έχει γίνει τώρα ένας βασικός στόχος για τους ερευνητέ μας, για τα πανεπιστήμια μας, για τα ερευνητικά μας κέντρα, διότι εκτός από το κύρος το να μπορέσει κανείς να φτάσει στην αριστεία ε, έχει ως αποτέλεσμα την ζωή πόρων ώστε να διατηρηθεί αυτή η πρωτοπορία. Οπότε γι' αυτό και μας ζητούν, επειδή είμαστε νομοθέτες, να ξεκαθαρίσουμε την έννοια αυτή και κυρίως να ξεκαθαριστεί το ε, πώς εκτιμάται, πώς, πώς μετράτε. Γι' αυτό και έχουμε εδώ προσκαλέσει όλους αυτούς τους ε, εμπειρογνώμονες και θα πρέπει μας να τους ρωτήσουμε πώς μετράτε η αριστεία, θα πρέπει να επιφυλάσσουμε αυτή την έννοια στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 ε, στις βασικές επιστήμες ή αυτό να αφορά και την ε, οικονομία, να αφορά και την ανταγωνιστικότητα ε, και επομένως είναι εδώ να μιλούμε για την δημιουργία γνώσης και ή και για το πώς η έννοια αυτή θα μεταλαμπαδευτεί και στην κοινωνία και στην αγορά και πώς θα μετρηθεί. Αυτό επομένως θα θέλαμε να το συζητήσουμε μαζί σας. Δηλαδή το πώς θα διευρυνθεί αυτή η έννοια. Και επομένως όσοι παρακολουθούν το έργο μας γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί παγίως. Γιατί οπωσδήποτε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι στο επίπεδο αυτό υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των μελών. Η δε κατάσταση αυτή είναι δυνατόν να μας οδηγήσει ε, σε ένα ρήγμα μεταξύ των κρατών μελών το οποίο ε, δεν είναι καλό. Επομένως εμείς θα πρέπει να ε, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε άριστοι, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την συμμετοχή. Γιατί έτσι πρόκειται να ωφεληθούμε ως Ευρωπαίοι. Πρέπει όμως να βρούμε τον πιο δόκιμο τρόπο. Και σε αυτό το πλαίσιο θα μιλήσουμε για έρευνα, για διακυβέρνηση και επίσης εις βάθος θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στους ανθρώπινους πόρους. Και εγώ δεν θα σταθώ μόνο ε, στις δράσεις ε, Κιουρί που όπως ε, θα θυμάστε όλοι έγιναν θα δούμε τι πρέπει όλοι να κάνουμε ούτω ώστε να ελκύσουμε τους καλύτερους από τους νέους μας σε μια σταδιοδρομία επιστημονική και τι θα κάνουμε ούτως ώστε να τους ε, κρατήσουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες ούτως ώστε να έχουν την επιθυμητή κινητικότητα και να δούμε τι άλλα μέτρα μπορούμε να λάβουμε ούτως ώστε να προχωρήσουμε προς τον τελικό στόχο να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά και για τον ερευνητή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα εκατομμύριο ερευνητέ. 3% του ΕΠ να αφιερώσουμε και επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για την έρευνα ούτω ώστε να έχουμε έναν πυλώνα, τον πυλώνα της προστιθέμενης αξίας και έτσι να βελτιώσουμε την καινοτομία και ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας ε, πυλώνας που στην σημερινή οικονομική συγκυρία να μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε στην Ευρώπη να έχουμε βιωσιμότητα, να έχουμε απασχόληση, ποιότητα, να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στη μακροσμιοποίηση. Αυτό δεν είναι εύκολο. Είμαι όμως βέβαιη ότι με αυτά τα οποία τώρα θα ακούσουμε θα μας κατέβουν πάρα πολύ αξιόλογες ιδέες. Έχετε τη σκητάλη, Πρόεδρε, πάλι. Ευχαριστώ την κυρία Μαντουρέλ για την παρέμβασή της δώσουμε τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Ε, καταρχήν θα πάρει το λόγο ο κύριος ε, Μαριάνο Καγκό, ο οποίος ε, είναι πρωθυπουργός τεχνολογίας, επιστημών και ανάπτυξης εκπαίδευσης. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα πω δύο λόγια στα πορτογαλικά καταρχήν και κατόπιν θα μιλήσω στα αγγλικά. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ήτρε και ε, τους συζητητές αυτού του προγράμματος πλαισίου για την ευκαιρία που έχουμε να υλοποιήσουμε μια διευρυμένη συζήτηση για αυτό το θέμα και θα ήθελα ιδίως να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, ε, όλους όσους ε, υλοποιήσατε αυτό το πρόγραμμα. Εγώ ε, είχα το προνομίο να παρακολουθώ από την αρχή σχεδόν όλα τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξη στην Ευρώπη και μπορώ να σας πω ότι αυτό σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες προτάσεις που παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την απόψή μου. Ε, μέχρι σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τους ε, ηθήνοντες για όλο το έργο τους που πρέπει να ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να καταρθώσουμε να έχουμε αυτή την πρόταση ενωπιών μας. Λεχθέντος αυτού. Θα μιλήσω αγγλικά αν δεν σας πειράζει. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω χρειάζεται περαιτέρω οπτική αναπαράσταση το πρόγραμμα ορίζοντες για να καταλάβετε τι ακριβώς συζητάμε. Αλλά εφόσον έχετε τις διαφάνειες της παρουσίασής μου θα τις διτρέξω εν συντομία. Το πρώτο σημείο που ήθελα να θέξω ήταν το εξή. Ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή αρχή που θα πρέπει να αναθερεθεί προσεκτικά, αυτό προβλέπεται και τον κανονισμό, αλλά και που χρήζει κάποιων βασικών βελτιώσεων. Θα ήθελα να μιλήσω για την πρώτη ανάγνωση και μετά να τονίσω κάποιες ευκαιρίες οι οποίες ε, θα αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση της πολιτικής για την επιστήμη και τεχνολογία τα επόμενα χρόνια. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαβάσετε τις διαφάνειές μου στην οθόνη, αλλά θα έχετε και αντίγραφα. let, let να περάσω γρήγορα γρήγορα να σας παρουσιάσω ποια, έχει, ποια είναι η κατάσταση. Τα επόμενα χρόνια έως το 2020 εξετάζουμε. Θα τροποποιηθεί δραματικά η κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε και πλέον διαμορφώνεται στα 50, όχι συγγνώμη, προσθέθηκαν 50 εκατομμύρια φοιτητέ στα ήδη υφιστάμενα 100 εκατομμύρια των περασμένων ε, δεκαετιών. Και ο αριθμός των ερευνητών ακολούθησε την ίδια κατεύθυνση λοιπόν. Και στην περίοδο 2002 έως το 2007 ο αριθμός των ε, ερευνητών αυξήθηκε κατά 25% από 5,7 εκατομμύρια σε 7,1 εκατομμύρια ερευνητές κοιτώντας τις δημοσίευσεις τώρα και τον ρυθμό αύξησης των διεθνών τέτοιων δημοσιεύσεων από το 1 εκατομμύριο περάσαμε στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν λέω αυτό. Ο κόσμος μεταβάλλεται ταχύτατα προς το καλύτερο, προς το καλύτερο. Γιατί ασχολούνται όλο και πιο πολλοί άνθρωποι με τις ε, έρευνες και υπάρχουν και γίνονται όλο και πιο πολλές επενδύσεις και θα υπάρχουν όλο και πιο πολλές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια των ερευνών αυτών. Άρα, ανταποκρινόμενοι στο σενάριο αυτό, εξετάζουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη. Άρα, σημείο αφετηριασμού είναι ότι η έρευνα αποτελεί ε, κινητήριο δύναμη για τις αξίες και τις οικονομίες και για το πολιτικό προσκήνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Φυσικά θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις αλλαγές της παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης να δούμε τι γίνεται για τα θέματα οικονομικής και βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα ταλέντα που διαθέτουμε αλλά θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση και τους περιορισμούς της χρηματοδότησης σε όλη την Ευρωζώνη. Ωστόσο, και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει προσεκτικά να αναλύσει αυτή η πρόταση στον ορίζοντα 2020. Το θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας φαίνεται ότι έχασε κάποιον από τον αρχικό του ρόλο. Δεν είναι σαφές πως οι οικονομικοί περιορισμοί και οι πρακτικές της οικονομίας ε, αποτυπώνονται. Θεωρώ ότι δεν αποτυπώνονται καθόλου στην πρόταση και δεν δίδεται προτεραιότητα στην κατεπίγουσα ανάγκη να τονίσουμε και να προωθήσουμε, να ενισχύσουμε την ε, πολιτική, το πολιτικό εκλογικό κοινό προκειμένου ο κόσμος να απαντήσει προς τους πολιτικούς ότι ναι, θέλουμε προτεραιότητα στην έρευνα. Και η βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης δεν θεωρείται επαρκώς ως μια ευκαιρία. Άρα υπάρχει κάποιο περιθώριο λοιπόν στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο. Για να το θέσω σε πρακτικούς όρους τώρα. Αν ε, θα πρότεινα μία πρακτική προσέγγιση για τη βελτίωση των ορίζον, του ορίζοντα 2020 και νομίζω ότι αυτό κάνουμε στην παρούσα φάση, θα σχολίαζα κάποια παραδείγματα. Δεν πρόκειται για μία συστηματική προσέγγιση, πρόκειται για κάποια τυχαία παραδείγματα. Ενδεκτικά, μάλλον. Να σας τα αναφέρω. και θα εξετάσω λεπτομερώς κάποια για τις κοινωνικές ε, επιστήμες. Περιορίζεται ο ρόλος τους στο πρόγραμμα πλαίσιο και νομίζω ότι υπάρχει μια γενική συνένεση σε όλη την Ευρώπη και μεταξύ των ηθήνων ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ας φανταστούμε να χρησιμοποιείτε τέτοιο επιχείρημα για τις ε, επιστήμες πληροφορικής. Ότι, α, κοιτάξτε, αφού είναι παντού οι επιστήμες αυτές, θα χρειάζεται να τονιστούν ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ απαραίτητες για τα επόμενα χρόνια λόγω της αλλαγής των νομών της κοινωνίας σε όλη την Ευρώπη που θα πρέπει να γίνουν καλά κατανοητές. Το δεύτερο σημείο είναι η επιστήμη και η κοινωνία. Και αυτό έχει ελαχιστοποιηθεί ω προς τη σημασία του και είναι κρίσιμη η σημασία του για την ενίσχυση των ε, εκλογικών περιφερειών. Θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια, ακόμα και μετριοπαθή. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μετριοπαθή η προσπάθεια τη Ευρώπη στον τομέα αυτό, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέων ταλέντων, στην ανάπτυξη μιας ε, κοινή ε, κατανόηση ε, τη επιστήμη και στην πρόθεση τη γενικότερη συζήτηση. Για να περάσουμε τώρα στην έρευνα. Υπάρχει ένα παλιό ερώτημα, το οποίο ακόμα δεν έχει απαντηθεί όμω. Το πρόβλημα τη ε, εξαιρετική έρευνα σε όλα τα κράτη-μέλη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο στα προγράμματα πλαίσιο από την αρχή Πώς θα προωθηθεί λοιπόν η αριστεία στις ερευνές σε όλα τα κράτη-μέλη, σε πολύ μικρά κράτη-μέλη ή σε περιφέρειες αναπτυσσόμενες. Νομίζω ότι σχέδια όπως τα βραβεία για την αριστεία σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθηθούν. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια ελάχιστη χρηματοδότηση, αλλά να έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σαφώς και άλλες προτάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Κατά δεύτερον, συνεργασία στην έρευνα εντός των συνόρων. Για επιδοτήσεις δηλαδή, συνεργασίας ή μη συνεργασίας. Υφίσταται ένα πρόβλημα. Ως τώρα, στο έντομο πρόγραμμα πλαίσιο δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο για τέτοια έρευνα σε συνεργασία. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα διασυνοριακός. Έχει αναπτυχθεί αυτή η έρευνα συνεργασίας και τα προγράμματα FED ήταν πάρα πολύ σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά θεωρώ ότι είτε θα πρέπει να τονίσουμε εκ νέου το πρόγραμμα FED ή να δημιουργηθεί ένα νέο πρόγραμμα για το ERC, ένας νέος ρόλος για το ERC που θα προωθεί και την αριστεία αλλά και την συνεργασία. Και συγγνώμη που τρέχω, αλλά βιαζόμαστε. Ένα άλλο ζήτημα είναι η έρευνα συνεργασίας ως βάση για προηγμένη κατάρτιση στη βιομηχανία ή στον ακαδημαϊκό κόσμο. Η Marie Curie, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Marie είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά φαίνεται ότι έχει κολλήσει στην αρχική του, πρωτότυπη του μορφή. Δεν έχει λάβει υπόψη τις τεράστιες αλλαγές που έχουν προκύψει στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος πλαισίου δημιουργεί ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για την προηγμένη κατάρτιση των καλύτερων φοιτητών και θα ήταν μάλιστα καλός τρόπος προσέλκυσης φοιτητών από χώρες και οργανώσεις που δεν εμπλέκονται, δεν συμμετέχουν σε πολλούς τομείς ε, ε, ερευνών, για παράδειγμα σε βιομηχανικούς τομείς. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την έρευνα εργασία και τη χρηματοδότηση την ευρωπαϊκή ως βάση για την κατάρτιση αυτή την προηγουμένη, θεωρώ ότι αποτελεί μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να δράξουμε. Και τώρα γρήγορα γρήγορα να σας αναφέρω κανένα δύο σημεία. Ένα αφαιρετικό σημείο το οποίο αισθάνομαι όμως υποχρεωμένος να αναφέρω. Δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα στην αίθουσα Φιλιπ αλλά θεωρώ ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας θα πρέπει να αναπτυχθεί. Είναι μία καλή αρχή η οποία όμως πρέπει πλέον να αναθεωρηθεί. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκός Χώρος ε, έρευνας δεν αποτελεί έκφραση της ευρωπαϊκής κοινή αγοράς στον τομέα της έρευνας, γιατί αυτό αποτελεί μία συχνή ε, παρανόηση γιατί η κινητικότητα, η διακίνηση των ιδεών ήταν αυτή που προετοίμασε το, την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Άρα υποβαθμίστηκε πλέον ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ερευνών. Δεν αναγνωρίζεται πλέον και ο κόσμος αναφέρει πλέον ότι πρέπει να πετύχουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ερευνών. Όχι, όχι. Πρόκειται για ένα σύστημα όλων των εταίρων, όλων των οργανώσεων, όλων των φορέων. Θα πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτός ο στατικός ορισμός του χώρου, να το αποκαλέσουμε φιλοδοξία, δράση. Υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις που συνάδουν με αυτό το A του ERA για να αλλάξουμε τον ευρωπαϊκό χώρο ερευνών και βλέπω ότι πρέπει να περάσω στα συμπεράσματά μου. Ε, ένα άλλο παράδειγμα. Ένα άλλο θέμα είναι τα βλαστοκύτταρα. Ένα τομέα ο οποίος σχετίζεται με την επιστήμη γιατί μυρίζει θείο, σαν το διάβολο. Αλλά ως επιστήμον θεωρώ ότι είναι περίεργο να κοιτάω το άρθρο 16. Εδώ βλέπετε ένα αντίγραφο του άρθρου 16 που τονίζει με κόκκινους χαρακτήρες τη σημασία, τη δραματική σημασία των ε, βλαστοκυτάρων. Τα εμβριονικά βλαστοκύτταρα είτε τα χρειαζόμαστε είτε όχι αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει έρευνα είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή είναι η επιλογή που θα κληθείτε ως πολιτική να λάβετε. Υπάρχουν άλλες δύο ευκαιρίες στις οποίες δεν έχουμε απευθυνθεί. Το διάστημα, πρόεδρε, σας παρακαλώ ένα λεπτό αν θέλετε να μου δώσετε. Ξέρω ότι ένα από τα μέλη μας έχει κολλήσει και δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι στη Σαουδική Αραβία. Άρα έχουμε ο καθένας τρία λεπτά παραπάνω. Στο διάστημα λοιπόν. Το διάστημα ασφαλώς και είναι κρίσιμο για την οικονομική ανάκαμψη στο παγκόσμιο επίπεδο αλλά και για την Ευρώπη ιδιαίτερος. Θεωρώ ότι η πρόταση ορίζων 2020 δεν είναι ε, δεν αποτυπώνει την αναγκαία διαίρεση των αρμοδοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, για το διάστημα. Τώρα, η βιοιατρική. Δεν μπορούμε να κοιτάμε στη βιοιατρική τα μεμονωμένα μόνο έργα γιατί χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη οργάνωση, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, μακροπρόθεσμα έργα. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι τεράστια η πολιτική σημασία του τομέα αυτό. Τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι η ειρήνη. Και με αυτό κλείνω, Πρόεδρε, κλείνω με την ειρήνη. είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι και Αιγύπτιοι επιστήμονες συνεργάζονται από κοινού. Πολλοί συνδράμουν στο έργο αυτό, όχι όμως η Ευρώπη. Και θα ήθελα το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 ε, να συνδράμει σε, αυτή, σε αυτό το εγχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ε, κύριο καθηγητή για την παρέμβασή του. Θέλω ε, να ξεκαθαρίσω ότι, κοιτάξτε, όταν μακρηγορείτε, αφαιρείτε το χρόνο από άλλους συζητητές και δεν είναι αλήθεια ότι κάποιος λείπει, γιατί αντικαταστάθηκε έτσι, λοιπόν. Ο χρόνος παραμένει όπως είχε προγραμματιστεί και τα τρία λεπτά συσσωρεύονται στο χρονοδιάγραμμα της ακρόασης. Δεν είναι κακία λοιπόν από την πλευρά της Προεδρίας, απλώς πρόκειται για μια απόπειρα να έχουμε μια καλά οργανωμένη συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο καθηγητή Κάκου. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Κούρτ Ντεκελατέρ, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας για την Λίγκα των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή που κάλεσε τελικά των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Πανεπιστημίων εδώ σήμερα το πρωί για να σχολιάσει επί της, προτάσ... επί της πρότασης για τον ορίζοντα 2020. Θεωρώ ότι τα μέλη της ΙΤΡΕ μέχρι τώρα γνωρίζουν ε, τι είναι το ΛΥΡΟΥ. Πρόκειται για τη λύκη 21 ερευνητικών πανεπιστημίων ε, από την Ευρώπη, από ένα χώρε και καθημερινά προσπαθούμε να προωθήσουμε ε, τα συμφέροντα της έρευνας στην Ευρώπη. Θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο. Έχω δέκα σημεία που θέλω να αναφέρω και θέλω να αφιερώσω ένα ε, λεπτό σε κάθε θέμα. Ε, δεν ε, υπάρχουν διαφάνειες, έτσι λοιπόν απλώς θα πρέπει να με ακούσετε. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα 15 λεπτά ίσως ε, θα πρέπει να δούμε τις προτάσεις όπως έχουν κατατεθεί από την Κομισιόν και επίσης έχω στη σχολιά μου συμπεριλάβει ένα πρώτο συνδεσμό με το έγγραφο εργασίας που δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη εκπονούν τις τελευταίες εβδομάδες ε, το γραφείο ε, για, ε, για ορίζοντα 2020 από την κυρία Μαντουρέλ και το έγγραφο για τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του κυρίου Έλερ. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιους συνδέσμους και με τα δύο έγγραφα κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Θα διαρρέσω την παρουσίασή μου σε δύο κυρία μέρη. Καταρχήν, θα ήθελα να πω στους κυρίους βουλευτές, θα αναφέρω πέντε σημεία, επί των οποίων ε, θέλω να σας ζητήσω να μην τροποποιήσετε τις προτάσεις της Κομισιόν. Και σε ένα δεύτερο μέρος θα ήθελα να αναφέρω πέντε σημεία, επί των οποίων ε, θα ήθελα να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά για να δείτε αν μπορούν να διατυπαθούν καλύτερα από αυτό που έχουμε σήμερα επιτάπητος. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα πέντε σημεία επί των οποίων θα ήθελα εσείς ε, να μην τροποποιήσετε τίποτα. Καταρχήν, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι η επιστημονική αριστεία διατυπώνεται ως ε, το πρωταρχικό κριτήριο χρηματοδότησης υπό τον ορίζοντα 2020. Θα θέλαμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτή την αρχή και επανέρχομαι στις εισαγωγικές ε, δηλώσεις της κυρίας Μαντουρέλ όταν ε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι προφανώς ε, ε, όλες οι χώρες ε, της Ευρώπης δεν είναι το ίδιο επιτυχημένες ε, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και βέβαια το ΛΕΡ προσφέρει συνεργασία σε ό,τι αφορά τις αποκαλούμενες δραστηριότητες γεφύρωσης που προτείνονται στα έγγραφα της Κομισιόν στον τομέα της έρευνας όπως και στον τομέα της διαφορετικής περιφερειακής πολιτικής. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες που στερούν και να οικοδομήσουν ικανότητα έρευνα, αλλά η χρηματοδότηση πρέπει να γίνει μέσω των διαφορετικών ταμείων ή άλλων πηγών πέραν του ορίζοντος 2020. Ε, το δεύτερο σημείο με το οποίο είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και θέλουμε να διατηρήσουμε ως έχει είναι το ποσοστό αποζημίωσης του άμεσου κόστους 100% με 20% αποζημίωση του έμεσου κόστους. Ξέρουμε ότι κυκλοφορούν διάφορα μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν για μας ως πανεπιστήμια να ε, χορηγήσουν περισσότερα χρήματα, αλλά προτιμούμε να διατηρήσουμε το 100% και το 20% την προσέγγιση αυτή, γιατί η διαχείριση όλων των project θα είναι πιο απλή με τον τρόπο αυτό, θα σεβόμαστε καλύτερα τους κανόνες, ε, εθνικούς κανόνες χρηματοδότησης και τα πανεπιστήμια θα μπορούν να προσελκύσουν ε, προσωπικό που να εργάζεται αποκλειστικά για τα έργα του ορίζοντος 2020. Θα ήθελα να πω παρόλα αυτά ότι ο κανόνας 100% 20% είναι το ε, απολύτως ελάχιστο. Οτιδήποτε κάτι από αυτό θα θέσει σε κίνδυνο ε, την ε, συμμετοχή των πανεπιστημίων στην Ευρώπη στο πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 γιατί για μα η βιωσιμότητα της έρευνα είναι κάτι θεμελιώδε. Δεν μπορούμε λοιπόν πλέον ε, να συμμετάσχουμε σε χρηματοδότηση έρευνα που να μην οδηγεί σε μια υφόρο κατάσταση για τα πανεπιστήμια. Προφανώς ε, δεν θα είμαστε αντίθετες σε μια αύξηση ε, της αποζημίωσης ε, για τις άμεσες, δαπα... άμεσες δαπάνες, όμως πρέπει να σας πω ότι το 20% είναι το απολύτως ελάχιστο για αυτές τις άμεσες δαπάνες. Επίσης, θα ήθελα να χαιρετήσω το γεγονό ότι ο ΦΠΑ επίσης θα είναι επιλέξιμο κόστος, επιλέξιμη δαπάνη στο μέλλον. Ήταν πρόβλημα αυτό για πολλά πανεπιστήμια, δηλαδή ότι δεν επιστρεφόταν ο ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν αυτό είναι είναι ένα πολύ καλό σημείο στις προτάσεις. Και τέλος, ε, θα ήθελα να διασφαλίσω ότι δεν, υπάρχει, δεν θα υπάρχει σύγχυση στο μέλλον σε ό,τι αφορά τα project που θα χρηματοδοτούνται μόνο για 70%. Ε, ίσως ε, θα πρέπει εδώ να απευθυνθούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένας σαφής ορισμός για την καινοτομία και για το ποια project στον τομέα της καινοτομίας οδηγούν μόνο ε, σε ε, αποζημίωση της, του 70%. Ένα ακόμη σημείο που θέλω να θίξω είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές τις ερευνητικές. Είμαστε ικανοποιημένοι που αναπτύσσονται οι υποδομές για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό φυσικά είναι αυτονόητο, αλλά εδώ είμαστε κάπως όφρονες. Πρέπει να είναι και σε ότι οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές ε, δεν θα πρέπει ε, να είναι το κυρίαρχο κόστος του προπολογισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνα. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί καλή διαχείριση, σωστή έλεγχη, αναθεώρηση και θα έλεγα ότι μία σειρά των υποδομών αυτών μπορούν να έχουν μόνο προσωρινό χαρακτήρα, έτσι λοιπόν να μην συστήνονται υποδομές με την ιδέα ότι θα είναι διαβίου. Ένα ακόμη σημείο που θέλω να προσθέσω στο θετικό κατάλογο είναι η επιβεβαίωση της θέσης του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου Ηλίρου. Ε, ήταν ε, ε, μεγάλος χρηματοδότης ε, του ERC, εκπροσωπούμαστε με 21 πανεπιστήμια, εκπροσωπούμε πάνω από 20% ε, όλων όσων λαμβάνουν επιδοτήσεις. Έτσι λοιπόν για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσο στη συνολική πολιτική της έρευνας. Παρόλα αυτά ε, υπήρξε κάποια έπληξη για το συνολικό ενθουσιασμό για τον προπολογισμό του ERC του Ερευνητικού Συμβουλίου. Κατά την άποψή μας θα χρειαστεί ακόμη ψηλότερο κονδύλι για το ERC, γιατί αν δείτε τώρα τα αριθμητικά στοιχεία θα παρουσιαστεί μείωση του προπολογισμού όταν θα ολοκληρωθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και θα ξεκινήσει ορίζοντας 2020. Το 2013 το ERC σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία θα έχει προπολογισμό 1,8 δισεκατομμύρια και το 2014 1,6 δισεκατομμύρια μόνο. Έτσι λοιπόν αυτό δεν είναι κάτι θετικό. Και δεύτερον πιστεύουμε ότι λαμβάνοντα υπόψη ε, την ε, επιτυχία των εφαρμογών ε, των επιδοτήσεων, η ERC ότι ένα αυξημένο προπολογισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο ποσοστό επιτυχία όλων των αιτήσεων του ERC. Ένα πέμπτο σημείο που θέλω να θέσω στο θετικό κατάλογο είναι τα πολλά μέτρα που στοχεύουν στην απλούστευση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με όσα διατυπώνονται στο σχέδιο κειμένου για την συμμετοχή, για το streamlining των κοινών κανόνων, την ευθυγράμμιση των κοινών κανόνων για όλα τα τμήματα του προγράμματος και για όλους τους πρωταγωνιστές, του γεγονό ότι δεν υπάρχει πλέον απέτηση να ε, υπάρχουν time sheets ε, για όσους εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και επίσης είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την συνεχή αύξηση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών σημείων, με τη λογοδοσία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά σημεία και θέλω να πω ότι οι συγητές επίσης το τόνισαν αυτό και κυρίως ο κύριος Έλερ ε, πολύ σωστά λέει ότι πρέπει να υπάρχει η καλή ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης, της ευελιξίας, ε, της αξιοπιστίας και της λογοδοσίας. Αυτά όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά να φτάσω τώρα στο δεύτερο κατάλογο των πέντε σημείων. Όπου εδώ θέλουμε να ζητήσουμε μια αναθεώρηση κατά κάποιο τρόπο ή τουλάχιστον καλύτερη διατύπωση του σημερινού κειμένου. Καταρχήν, έχουμε τον προπολογισμό για τις δράσεις Marie Curie ε, και για τις δεξιότητες στην κατάρτιση και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Απογοητευτήκαμε ιδιαίτερα από τα κονδύλια που κατανέμονται στις δράσεις Marie Curie, γιατί αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία θα μειωθεί ο προπολογισμό από ένα δισεκατομμύριο σχεδόν στο 2013 στα 0,7 δισεκατομμύρια το 2014 και θα φτάσει το επίπεδο το 2013 μόνο το 2019. Έτσι λοιπόν, ε, όπως ξέρετε, ήταν μεγάλη απογοήτευση γιατί το Marie Curie ήταν ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα μέχρι τώρα και ενίσχυσε την ποιότητα και την αριστεία του επιστημονικού προσωπικού με ένα πολύ σημαντικό τρόπο. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να το ξανασκεφτούμε το ζήτημα. Και επίσης εδώ στα κείμενα που έχουμε επιτάπητος θα πρέπει να γίνει σαφή σύνδεσμος με όλα όσα εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της εφαρμογής ή των μνημονίων εφαρμογής που εξετάζουμε με την Επίτροπο σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Είναι σαφές ότι οι προτάσεις της Κομισιόν στο παρελθόν για τη χάρτα και για το κωδικά και για το λογότυπο, για τις στρατηγικές ε, γνώσεις και ανάπτυξη είναι πολύ θετικά σημεία και οι αρχές που αναπτύχθηκαν από την Κομισιόν για την ε, διδακτορική κατάργηση, για το φύλλο, ε, είναι πρωτοβουλίες ιδιαίτερα αξιόλογε και ίσως μπορεί να γίνει ένα σαφή σύνδεσμος εδώ με αυτά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αφιερώνεται επαρκή προσοχή στις δεξιότητες, στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη της διαδρομίας. Ένα δεύτερο σημείο για το οποίο, το θέλω να, στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι ότι θα θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη διαβεβαίωση περισσότερων πρωτοβουλειών από κάτω προς τα πάνω στον τομέα της έρευνας, στην προτεραιότητα 2 και 3 του προγράμματος, ε, δηλαδή για την ε, ε προκλήσεις ε, τις κοινωνικές και την ηγετική θέση στον τομέα της βιομηχανίας. Η βασική έρευνα ε, συνήθως ε, γίνεται από πάνω προς τα κάτω. Εμείς θέλουμε όμως το αντίστροφο και θέλουμε να το διασφαλίσουμε αυτό στα περισσότερα τμήματα του προγράμματος. Ε, το είπε αυτό το προηγούμενο ομιλητή ότι, με ε, ε, ότι υπάρχει επέκταση του συστήματο των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών. Ε, ΦΕΤ, όμω, εμεί ελπίζουμε ότι θα ενταχθούν σε πιο προσανατολισμένα προγράμματα και όχι μόνο στην προτεραιότητα 1. Έτσι, λοιπόν, θα έλεγα ότι ο προπολογισμό ΦΕΤ θα πρέπει να ε, καταναμηθεί σε όλα τα προγράμματα και όχι να περιορίζεται μόνο στην πρώτη προτεραιότητα και ε, πιθανότατα. Ε, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ χαμηλός ο προπολογισμός έτσι όπως έχει διατυπωθεί αυτή τη στιγμή. Τώρα εδώ ε, θέλω να συνδεθώ και με, προηγούμενο, με τον προηγούμενο μιλητή αλλά και με όσα αναφέρθηκαν από τους εισηγητές ότι θα θέλαμε να δούμε μία πιο ορυτή διαβεβαίωση για την έρευνα στις ε, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Η Επιτροπός ήταν πολύ σαφής για την υποστήριξή της για τις ε, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες ε, στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είναι πρόβλημα να το αναφέρουμε αυτό πιο ρητά στο κείμενο. Από την άλλη, Επίσης, θα ενεργοποιήσουμε και τα δικά μας μέλη των επιστήμιων να σταματήσουν να παραπονιούνται συνεχώς για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης, θα πρέπει να ανοίξουν και σε άλλους τομείς και στη μηχανική, στην ιατρική και πρέπει επίση να αρχίσουμε να εργαζόμαστε με έναν πολυτομιακό τρόπο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Κομισιόν επίσης μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα το τονίσει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τέταρτο σημείο. Στον κατάλογο είναι το θέμα της ε, αποζημίωσης ε, του κόστους ε, που θα βασίζεται σε πλήρη, σε πλήρη οικονομική αξιολόγηση του κόστους εδώ. θα ήθελα να σας πω τη Λύρου, πάρα πολύ καιρό εργάζεται για το θέμα αυτό και απογοητεύτομαι που ε, η πλήρης ετοιμολόγηση αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα του full costing. Κατάλαβα ότι κάποιοι από την δελτά προπολογισμού είχαν πρόβλημα με αυτό ότι δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη επλούστευση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ. Δεν μιλάμε μόνο εδώ για επιστροφή δαπανών σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, όμως για το πανεπιστήμια αυτό αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο εργαλείο εσωτερικής διαχείρισης. Πρέπει να ξέρετε ότι όλα σε κάνουμε ως πανεπιστήμια κοστίζει. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν δεν μπορεί αυτό να συμπεριληφθεί ως ένα σύστημα αποζημίωσης, επιστροφής των δαπανών, τουλάχιστον θα πρέπει να αποτελεί μια οικονομική διαχείριση, για μια οικονομική αρχή για την εσωτερική διαχείριση των πανεπιστημίων. Και ένα ακόμη σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το άρθρα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε ό,τι αφορά στα άρθρα αυτά, ανησυχούμε κάπως ότι δημιουργείται ανισορροπία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Αν ε, δούμε τα άρθρα που έχουν να κάνουν ε, με τον ορισμό των λογικών συνδικών, αν δούμε την ε, αυξημένη έμφαση που δίνεται στην θέση σε εμπορία και στους των αποτελεσμάτων, αν δούμε και την πρόσβαση για την εκμετάλλευση, βλέπω εδώ μία ανισορροπία μεταξύ της των θέσεων των πανεπιστημίων και των θέσεων της βιομηχανίας. Θα πρότεινα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μια πιο ισορροπημένη διατύπωση για τα άρθρα αυτά, έτσι ώστε να εγγυηθούμε ότι και τα πανεπιστήμια και η βιομηχανία είναι ισότιμοι εταίροι σε κάθε σύστημα συνεργασία. που μπορεί να συσταθεί. Αυτά είναι λοιπόν τα 10 σημεία που θέλω να φέρω. Πέντε θετικά, πέντε επί των οποίων σα ζητώ να προσδώσετε μεγαλύτερη προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Και τώρα. Αντί του κυρίου Ταμάγιο, ο οποίος πρόκειται να έρθει, θα έρθει ο κύριος Χόρχε Βελάσκο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Ισπανικού Εθνικού Ερευνητικού Ιδρύματος. Κύριε Βελάσκο, έχετε το λόγο. Καλημέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, ακριβώς όπως ακούσατε, θα ήθελα να με συγχωρήσετε. Ε, μάλλον συγχωρήσετε τον διευθυντή μας, τον Πρόεδρο τα Μάγιο, για λόγους με καιρού δεν μπορούσε να είναι εδώ. Ε, όπως είπε ο παλιός φίλος, Ζωζέ Μαριάνο Γκάγκο, λόγω κάποιας αμοθίελας δεν μπόρεσε να πετάξει ο διευθυντής. Πάντως με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ και θέλω να σας πω ότι στο ΣΕΡΝ έχω προσπαθήσει να πετύχω κάποια πράγματα με τον ε, Ζωζέ. Και επομένω ε, εξοικειωθήκαμε από τότε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κυρίες και κύριοι, πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω ε, σας την ε, Επιτροπή ε, Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για το τι θα γίνει όσον αφορά το πρόγραμμα Horizon 2020 για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την επιστημονική αριστεία. Και θα ξεκινήσω με μια σύντομη παρουσίαση για ε, αυτά τα οποία ε, θέλω να σας πω τι έχει πει ο πρόεδρος ε, Ταμαγιο. Ακριβώς έγραψε τα εξή. Θα κάνουμε αυτή την σύντομη παρουσίαση για μέρος του, του του Ιδρύματός μας που ξεκινούμε από τη βασική έρευνα και φτάνουμε μέχρι την ε, μεταφορά της, ε, στο, στον τομέα της παραγωγής και οπότε τώρα έχουμε 15.000 ε, που εργάζονται για αυτό το σκοπό. Έχουμε 100 επίσης ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται μαζί μας και βρίσκονται σε όλη την Ισπανία και το Θεσία έχει 6% του προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη στην Ισπανία και επίσης έχουμε το 20% της επιστημονικής εθνικής παραγωγής και το 25% όσον αφορά ε, της ε, ευρεσιτεχνίας. Ε, έχουμε σημαντικά έργα υποδομής, έχουμε βιβλιοθήκες σε, σε δίκτυο σε όλη τη χώρα και έχουμε επίσης πάρα πολλά μεικτά κέντρα έρευνας και συνεργαζόμαστε με πανεπιστήμια και με άλλα νομικά πρόσωπα κρατικά και ιδιωτικά ισπανικά και στο εξωτερικό. Έχουμε οκτώ ε, τομείς ε, επιστημονικούς στους οποίους ε, εργαζόμαστε και επίσης αφορά όλες τις επιστήμες η δουλειά μας. Σε αυτή μας την πορεία με στον χρόνο παρακολουθούμε και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και επομένως φτάνουμε στο 30% όσον αφορά την επιτυχία για τις σχετικές προτάσεις. Τώρα έχουμε 400 project τα οποία χρηματοδοτούν στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου και έτσι έχουμε αισιοδοξία όσον αφορά το ότι πρόκειται να ξεπεράσουμε τα επιτεύγματα του προηγουμένου προγράμματος πλαισίου και έτσι θα ε, συνεχίσουμε και έτσι θα, να, να, να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά τους καλύτερους μαθητές στην Ευρώπη και συνεργαζόμαστε με τα θεσμικά όργανα όσον αφορά τον προγραμματισμό, την, πολιτική έρευνα και επίσης συμμεριζόμαστε τα μέσα πολιτικής της Ευρώπης και έτσι προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει και με τα μέλλοντα προγράμματα πλαίσια και γι' αυτό ε, συνεργαζόμαστε και με ε, εθνικά και ευρωπαϊκά ε, ιδρύματα και, και, και ομίλους νομικών προσώπων και εταιρείων. Επίσης, παρακολουθούμε την καινοτομία για να πετύχουμε τους στόχους που έχει τάξει η πολιτική Ευρώπη 2020. Όπως τα γνωρίζετε ε, και εσείς που συζητείτε εδώ το τι θα γίνει με το ορίζοντα 2020. Στις 30 Ενδεκάτου του 2011 δημοσίευσε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή όσον αφορά την ε, έρευνα και καινοτομία και αναμφίβολα πρόκειται για βήμα προς τα εμπρός, ούτως ώστε να μπορέσουμε ε, τη γνώση που έχουμε πετύχει να την μεταλαμβαδεύσουμε στην κοινωνία, ούτω ώστε να εστιάσουμε προσοχή μα όσον αφορά την καινοτομία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια ρητσική αλλαγή σε σχέση με το τι ίσχυε στο παρελθόν. Το θέση θεωρεί ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί με αυτή τη νέα πρωτοβουλία για να μην φτάσουμε ε, υποβάθμιση της ε, ποιότητας της έρευνας. γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση πρόκειται να βελτιώσει το τοπίο το οποίο ισχύει σήμερα στην έρευνα και έτσι θα έχουμε καλύτερη προσβασιμότητα ε, και για επιχειρήσει και για ερευνητέ. Θεωρούμε πάντω ότι στην πρόταση υπάρχουν κάποιε ακραίε θέσει. Θα πρέπει να δούμε τι λεπτομέρειε των προτάσεων για να, να δούμε πώ θα γίνει η, ε, η εφαρμογή, τι προτεραιότητε θα τάξουμε. Πάντως, και ας μην το συζητούμε σήμερα, ε, θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για την ε, χρηματοδότηση σε σχέση με την συμμετοχή στο πρόγραμμα 2020. Εμείς συμφωνούμε 100% ότι το σύστημα επιστροφής των εξόδων για το 7ο πρόγραμμα θα πρέπει να απλωστευτεί. Παρ' όλα αυτά, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν μοναδικό μοντέλο ε, αυτό το, το σύστημα ούτως ώστε ε, κατά αυτόν τον τρόπο πλήσονται κάποια ερευνητικά ιδρύματα τα οποία πρόσφατα έχουν πετύχει μια εξυγίανση των οικονομικών τους, συρρήγνωση των πραγματικών δαπανών ακριβώς όπως θέλει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, όμως ε, οι ενισχύσεις τώρα θα συρρήγνωθούν από πλευρά της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν, επομένως στον βωμό της απλούστευσης να περικόψουμε τόσο πολύ τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους που μας βοηθούν για αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Ε, φαντάζομαι ότι και οι άλλοι θα σας τα πούν που θα συμμετέχουν στα πάνελ. Τρεις προτεραιότητες έχουμε. Πρώτα-πρώτα έχουμε την ε, επιστημονική αριστεία που είναι το θέμα μας. Χρειάζεται τέτοια ποιότητα, ούτω ώστε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε τις δραστηριότητε μας που οι δραστηριότητες θεωρούμε ότι είναι συμπληρωματικές. Οπότε έτσι θα βοηθήσουμε όλη την επιστημονική κοινότητα, το Επιστημονικό Συμβούλιο, αναδιόμενες ε, δράσεις, ε, έρευνα, το, το Μαρία Κιουρί. Οπότε, σε αυτά τα πέντε πρώτα χρόνια πετύχαμε πάρα πολλά. Και επομένως θα πρέπει να πάμε στην ίδια και θα πρέπει να δούμε ότι οι νέοι ερευνητές βοήθησαν, υλοποιήθηκε το όραμα. Να έχουμε επομένως πάρα πολύ εξαιρετική ποιότητα σε αυτά που κάνουμε. Και επομένως πρόκειται για κάποιους οι οποίοι ε, ως ερευνητές άνοιξαν το δρόμο και θα τον ανοίξουν για τις επόμενες γενιές. Η επιλέξιμη αυτό το πρόγραμμα είναι επιστήμονες βραβευμένοι. Όμως, επίσης, ε, τους έχει μοναμηθεί σε κάποιους και το Νόμπελ. Τώρα, σε σχέση με το ε, όραμα αυτό, θέλουμε ε, όλοι με ανεξαρτησία να δουλεύουν για την έρευνα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε με αυτήν την αριστεία να είμαστε πρωταγωνιστές σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι προεκοδότηση θα υπάρξει. Έχουμε αυτά τα 15 δις. Θεωρούμε ότι για αυτά τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε στα πλαίσια του Μαρικιουρί δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα. Γιατί έτσι χιλιάδες νέων μπόρεσαν να ξεκινήσουν και να δρομολογήσουν μια επιστημονική σταδιοδρομία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα, αλλά έτσι προλιάνουμε το έδαφος και οι νέοι μπορούν να προχωρήσουν σε κάποια ριζοσπαστικά ε, προγράμματα και projects Οπότε θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο φιλόδοξοι. Θα πρέπει έτσι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την σταδιοδρομία του Ευρωπαίου ερευνητή. Να είμαστε μας αποτελεσματικοί και θα πρέπει να δούμε τι προϋπολογισμός θα υπάρξει και να έχουμε κάποια αύξηση σε σχέση με το, τη σημερινή προοικοδότηση. Βεβαίω να λάβουμε υπόψη τι οικονομικέ δυσκολίε των εθνικών ελληνικών ιδρυμάτων και έτσι να δούμε τι θα γίνει με τους ερευνητέ των διαφορετικών ε, χωρών και προσοχή να μην έχουμε ε, σημεία απόφραξης τα οποία να στραγγαλίσουν την επιστημονική διαδρομή των νέων ερευνητών. Οπότε θεωρούμε ότι τα προγράμματα κινητικότητας επίσης μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν ελκυστική μια επιστημονική σταδιοδρομία και έτσι να εξασφαλίσουν ε, πάρα πολύ καλούς, καλές, καλούς όρους για τους ερευνητές. Και επίσης το International Outgoing Fellowships ήταν κάτι το οποίο βοηθούσε αλλά δυστυχώς καταργήθηκε ούτως ώστε να μπορούν να πάνε σε χώρες που έχουν προχωρήσει πολύ οι νέοι επιστήμονες και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι κοινό πανομαστή στου τρεις πυλώνε είναι ε, μια πρωτοβουλία η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά όσον αφορά την επικοινωνία την πληροφόρηση και ε, είναι πάρα πολύ καλή η σχέση κόστους-οφέλους και γι' αυτό πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει ε, τα ίδια και στην επιστημονική έρευνα. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια διεπιστημονική ε, συμμετοχή και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να έχουμε έναν ε, οριζόντιο χαρακτήρα σε όλα αυτά ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτές τις Fed flagships και γι' αυτό το λόγο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στο πώς θα προχωρήσουμε για την, στην καινοτομία. Τώρα, στο τέταρτο σημείο αυτό που θέλω να σας πω, θα δούμε τι θα κάνουμε με τις υποδομές στην Ευρώπη. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα έχουμε ε, πρόοδο. Να πετύχουμε πρόοδο γιατί είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο ε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πώς η Ευρωπαϊκή Κλίμακα θα θα κάνει αυτά που θεωρούνται βασικά σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα εξή δύο. Πρώτα-πρώτα, συντονισμό με το, τα, Ταμείο Συνοχή και επίση να έχουμε. Ε, ε, να λάβουμε υπόψη τις, τις εθνικές υποδομές. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Επίσης, να σας πω τις τελευταίες μου σκέψεις ε, που είναι ε, προσωπικές αλλά νομίζω ότι ισχύουν για όλα αυτά τα οποία τώρα συζητούμε σήμερα όσον αφορά την ε, πολιτιστική, την σημερινή συγκυρία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι το οποίο ίσχυε από την αρχαιότητα. Θα πρέπει να έχουμε το, αυτό που λέμε ταλέντο, σύστημα αξιών και κάτι το οποίο ίσχυε από την αναγέννηση και κατά τον τρόπο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, έτσι, ε- έτσι έφτασε στο υψηλότερο σημείο της η ανθρώπινη δημιουργία και επομένως έχουμε κάποιες αρχές, κάποιες ε, αξίες οι οποίες δεν θα πρέπει να υποβαθμίζονται, να, να συσκοτίζονται από την σημερινή κρίση. Χρειάζεται δημιουργία, χρειάζεται ακαιρεότητα. Θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι ε, η επιστημονική πολιτική να λάβει υπόψη κάποια κριτήρια, κάποιες αρχές, κάποιους στόχους που αντιβαίνουν στην ιδεολογική βάση της σύγχρονης επιστήμης. στις επιστήμες που από όλα χρόνια ήταν κάτι στο οποίο αρίστευε η Ευρώπη. Τώρα δηλαδή δίνεται έμφαση στην καινοτομία και στην άμεση εφαρμογή της έρευνας. Χρειάζονται βέβαια κοινωνικο-οικονομικοί στόχοι, γιατί το δημόσιο χρήμα υποστηρίζει ε, την έρευνα ο φορολογούμενος και γι' αυτό και χρειάζεται να υπάρχει και υποχρέωση λογοδοσίας. Φοβάμαι πάντως ότι έτσι απομακρυνόμαστε από τις αρχές μας. Και προσοχή, γιατί το ήθετε ένα τώρα, η αριστεία η καινοτομία. Οπότε ξέρω ότι ως πρόεδρος του Συμβουλίου ε, αυτού για την έρευνα στην Ισπανία μας οδηγεί στο ότι θα πρέπει ε, να οδηγηθούμε σε κάποια κοινωνία και σε κάποια οικονομία οι οποίες να ωφελούνται από το έργο το οποίο εμείς επιτελούμε στο Ίδρυμά μας οπότε ε, θα ήθελα ε, λοιπόν όλες αυτές μας τις ιδέες να σας τις υποβάλω και έτσι νομίζω ότι με κοινέ προσπάθειες θα καταφέρουμε ε, το πρόγραμμα ορίζοντας 2020 να καταλήξει σε επιτυχία και έτσι να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο θέλουμε σε σχέση με τις ε, μεγάλες προκλήσεις που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε. Πάντοτε, επομένω, ε, και αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν μεγάλε αποφάσει και ελπίζουμε επομένω να καταφέρουμε να εξισορροπήσουμε του επιμέρου στόχου μα και να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστούμε τον κύριο Βελάσκο. Τώρα το λόγο έχει ο καθηγητής Πίτερ Γκρούς, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, του Max Planck Society της εταιρείας Max Planck ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να σας παρουσιάσω τις σκέψεις μας για το πρόγραμμα Horizon 2020. Ακούσαμε τρεις ομιλίες ήδη και χαίρομαι ιδιαίτερος ότι ακούγοντας τον Κέρτ Ντεκετελερή αλλά και του υπόλοιπου ομιλητέ, ουσιαστικά συμφωνούμε με τα δεκα σημεία τα οποία παρουσιάστηκαν. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι οι διοργανωτέ το α, αυτό, ανέμεναν αυτό και γι' αυτό λοιπόν μου έδωσαν ένα διαφορετικό ρόλο να απευθυνθώ και να απαντήσω τα τρία ερωτήματα. Γιατί χρειαζόμαστε ε, εξαιρετική βασική έρευνα στην Ευρώπη, ποια είναι η συνδρομή της, ε, του Ιδρύματος Max Planck σε ό,τι αφορά αυτή την εξαιρετική ε, επιστήμη και ποιε είναι οι θέσεις του Ιδρύματος Max Planck σε ό,τι αφορά ε, την ε, επιστήμη αυτή στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Τονίζω ουσιαστικά τα τέσσερα σημεία. Την γνώση, την εκπαίδευση, τα παγκόσμια προβλήματα και εδώ θα σταθώ για λίγο γιατί στο τέλος του αιώνα μας ο κόσμος θα έχει 10 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Ο κόσμος αυτός θα χρειάζεται πόρους. Έξι φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. 80% του πληθυσμού αυτού θα κατοικεί σε πόλεις. 42% θα είναι άνω των 65 χρόνων. Άρα σωστά αναθέτεται στους επιστήμονες να αντιμετωπίσουν αυτά τα παγκόσμια προβλήματα και αυτή, αυτό είναι το καθήκον μας. Να σας ε, πω γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον και από εμπορικής απόψεως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μακροοικονομία. Ο Ρόμπερτ Σόλο, βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ, κατέδειξε με σαφήνεια ότι οι νέες τεχνολογίες ευθύνονται για το 80% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ένας νέος ε, επιστήμονας, ο Hans Gersbach, απέδειξε ότι όσο πιο τεχνολογικά προηγμένη είναι μία χώρα, τόσο πιο πολύ αυξάνεται το ποσό των ε, βέλτιστων δαπανών σε βασική έρευνα. Άρα όσο πιο προηγμένη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο πολλά δαπανά σε τέτοια έρευνα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια μια προβολή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ε, σε παγκόσμιο επίπεδο της έρευνας και της ανάπτυξης. Και βλέπετε εδώ κάτι που θα σας κάνει να σκεφτείτε. Πάνω-πάνω βλέπετε τις Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι η χώρα με τι ε, πιο υψηλές δαπάνε. Θα ξέρετε ότι η Κίνα αυξάνεται ε, δραματικά εδώ. Έχει ξεπεράσει στις δαπάνε ε, την Ευρώπη και τις, δημοσιεύσει και βλέπετε κάτω-κάτω τις ευρωπαϊκές χώρες με την Γερμανία πάνω-πάνω αλλά με μια καμπύλη η οποία σε καμία περίπτωση δεν προσωμιάζει τις άλλες χώρες, τους βασικούς μας ανταγωνιστές ε, στη Δύση, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Αυτό λοιπόν για να μας υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τις ε, προδιαγραφές της συνθήκης της Λισαβόνας για το 3%. Ξέρετε το 2% θα πρέπει να προέλθει από τη βιομηχανία, αλλά και το 1% από τις δημόσιες ταπάνες θα πρέπει να δαπανάτε όντως, αν θέλουμε όντως να τονώσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Να σας δείξω ποιος είναι ο έμεσος αντίκτυπος σε, σε μακροοικονομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση α, της έρευνας και της ανάπτυξης. Βλέπετε μια μελέτη στις ΗΠΑ για τις ε, πατέντες, στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Βλέπετε λοιπόν σε όλες τις πατέντες ποια ήταν η πηγή της ε, γνώσης αυτής. 73% χρηματοδοτείται από δημόσιες οργανώσεις, από δημόσιους οργανισμούς. χρηματοδότηση στην καλύτερη μορφή της, σε μακροοικονομικό επίπεδο χρηματοδότηση. Ασφαλώς δεν μπορεί να προσμετρηθεί με αυστηρούς ε, ε νομισματικούς όρους, αλλά καταδεικνύει ότι χρειάζεται ε, τέτοια έρευνα που αποτελεί τη βάση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Να το πω αλλιώ, χωρίς δημόσια χρηματοδότηση δεν θα είχαν προκύψει αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αυτό ισχύει και ιδιαίτερα στην φαρμακοβιομηχανία. 80% των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προκύπτουν από δημόσια χρηματοδότηση στις χημικές πατέντες 75%, στους, στα ηλεκτρονικά 50%. Το συμπέρασμα το οποίο και βλέπετε εδώ, το πόρισμα της ε, μελέτης ε, από οικονομολόγο και πάλι που έχει αναλύσει όλα τα έγγραφα που αποτέλεσαν τη βάση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το πόρισμα λοιπόν είναι ότι οι κυβέρνησεις που ελπίζουν ότι η έρευνα που χρηματοδοτούν θα προωθήσει την κοινοτομία θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην αριστεία της έρευνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν αριστεία όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά και για την οικονομία. Επόμενο σημείο στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω. Ποια είναι η συνδρομή το Ιδρύματο μας Πλάνκ στην ε, αριστεία σε ό,τι αφορά την επιστήμη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ιδρύμα Μαξ Πλάνκ είναι μάλλον μικρός οργανισμός. Διευθύνει και διαχειρίζεται ερευνητικά κέντρα μεσαίου μεγέθους, περίπου 250 έως 500 υπάλληλοι κατά μέσο όρο. Βλέπετε λοιπόν μία μελέτη κοινωνιολόγων και ιστορικών που επικεντρώνονται σε θέματα δημιουργικότητα. Αυτό που βλέπετε στην σύνοψη είναι ότι η αριστεία στην επιστήμη προϋποθέτει αυτόνομες οργανώσεις. Στο πρόσφατο παρελθόν, και εδώ παραθέτω, ε, τα δημιουργικά μικρά κέντρα ήταν τα πιο δημιουργικά όπως το Πανεπιστήμιο Rockefeller και τα Ιδρύματα Max Planck. Τα Ιδρύματα λοιπόν αυτά του θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, αυτόνομα, αλλά να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Δεν μπορεί να είναι α, μόνα τους, χωρίς το ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό είμαστε λοιπόν στο εταιρεία Max Planck διαχειρίζεται περίπου 80 ιδρύματα. Έχουμε 16.900 απασχολούμενους και το ετήσιο ποσό χρηματοδότησής μας είναι 1,3 δισεκατομμύρια. Η αρχή αυτή είναι πολύ παρόμοια γιατί απασχολούμε πάντα τους άριστους σε κάθε τομέα και αν δεν υπάρχουν άριστοι δεν κάνουμε έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα. Βλέπετε ότι α, ...30% των διευθυντών μας είναι εκτός Γερμανίας, 88,6% των μεταδιδακτορικών μας είναι εκτός Γερμανίας και 46,7% των διδακτορικών φοιτητών μας είναι εκτός Γερμανίας. Στις φυσικές επιστήμες δε, η παραγωγή μπορεί να προσμετρηθεί βάσει ποσοστώσεων και βάσει αναφορών. Και βλέπετε ότι είναι η δεύτερη σε σημασία σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις εταιρεία μας. Έχουμε ιδρύματα κυρίως στη Γερμανία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δύο στην Ιταλία, ε, ένα στην Ολλανδία. Βρίσκεται σε φάση ίδρυσης ένα στο Λουξεμβούργο και χρηματοδοτείται, μάλλον η Φλόριδα έχει χρηματοδοτήσει άλλο ένα Ινστιτούτο. Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω, γιατί μπορεί να είναι σημαντικό για το θέμα το οποίο συζητήθηκε, ως προς το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε την αριστεία, στην αριστεία σε ε, χώρες που δεν έχουν καταφέρει να την πετύχουν. Να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο των Ιδρυμάτων Max Planck που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε θεσμική χρηματοδότηση με εταίρους από κάθε χώρα για πέντε χρόνια αρχική περίοδο ισχύω με την τα παράταση και να, σχημα... να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, όπως για παράδειγμα ε, σχολές κατάρτισης κτλ. Υπάρχει μία προϋπόθεση. Η χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσει τουλάχιστον κατά το ίμιση. Είναι πραγματικά υπέροχο το μοντέλο αυτό. Αν θέλετε λοιπόν να εισάγετε την αριστεία βάσει θεσμικής ε, χρηματοδότησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ήδη συγκεντρωθεί. Έχουμε για παράδειγμα ένα Ινστιτούτο, ένα Ινστιτούτο ε, στο Παρίσι με τις πολιτικές επιστήμες, ε, με το Κολέγιο του Λονδίνου, Επίσης, στην Ισπανία, επίσης ε, ε, προγραμματίζουμε να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι έγινε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να εξαγάγουμε και κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Οι συνεργασίες μας λοιπόν ξεκινούν από κάτω και κινούνται προς τα πάνω σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι ίσως δεν ε, διαβάζετε τους μικρούς χαρακτήρες ε, της ε, διαφάνειας. Βλέπετε εδώ λοιπόν στον πίνακα αυτό, στην τελευταία στήλη, ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ήταν πραγματικά καταλητική για την επιτυχία της εταιρείας Max Planck, γιατί υπήρχε σταθερή αύξηση από το πρόγραμμα πλαίσιο 4 έως 7 και πλέον έχουμε 6 δισεκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ε, χρηματοδότηση ανά έτος και πραγματικά είναι τεράστια αυτή η συνδρομή. Και δεν θα σας εκπλήξει αν σας αναφέρω από ποιο τμήμα του προγράμματος προέρχονται τα χρήματα αυτά. Το ERC όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, αποτέλεσε βασικό εργαλείο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση η ERC θα αυξηθεί, γιατί αν θέλουμε να προωθήσουμε την αριστεία, αυτό είναι το καλύτερο δυνατό εργαλείο για την εταιρεία Max Planck. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόγραμμα Marie Curie. Αν θέλετε να προωθήσετε την αριστεία, λέτε ότι θέλετε ένα εκατομμύριο παραπάνω επιστήμονες, πρέπει να προωθηθεί το πρόγραμμα Marie Curie, γιατί αυτό θα ενισχύσει την καριέρα των νεαρών επιστήμονων, ε, θα προωθήσει την κινητικότητα και θα βοηθήσει και τις χώρες που δεν έχουν αριστεί ακόμα στην επιστήμη. Επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλά project τα οποία δεν έχω χρόνο να σας παρουσιάσω. Η γύρανση αποτελεί ένα μόνο θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα γύρανσης για μία σειρά λόγων και στη γύρανση με υγιείς όρους. Αναφέρθηκε κάτι σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επιστήμες. Στον τομέα της ε, υγείας θα έχουμε την προσωπική ιατρική, την εξατομικευμένη ε, ιατρική. εσείς ως πολιτικοί θα πρέπει να φροντίσετε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την γενετική ανάλυση του καθενός μας. Τι θα γίνει με τα στοιχεία αυτή, θα μπορούν οι ασφάλειες να έχουν ε, πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Τι γίνεται. Πρόκειται για πράγματα τα οποία σε 10-15 χρόνια θα είναι πραγματικά πάρα πολύ κοινά και θα παίρνουν 10-15 λεπτά. Άρα τα πορίσματα θα πρέπει να διαφτηρίσουμε το ERC, θα πρέπει να κρατήσουμε την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, θα πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να βελτιώσουμε και την παγκοσμιοποίηση των προγραμμάτων. Σε ένα σημείο τονίζω εδώ πέρα με πράσινο χρώμα. Νομίζω ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου για την ε, εισαγωγή θεσμικής χρηματοδότησης ε, με ευέλικτο τρόπο είναι θετική. Νομίζω ότι η εταιρεία Max Planck μπορεί να βοηθήσει να ιδρυθούν τέτοια ε, ιδρύματα σε χώρες όπου δεν υφίστανται ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Γκρούς. Να ξεκινήσουμε αμέσω τη συζήτηση. Δύο λεπτά, να παρέμβαση, γιατί έχουμε καθυστερήσει, όπως γνωρίζετε. Η κυρία Χέντζοκ είναι η πρώτη που έχει στήσει το λόγο. Ε, ε, thanks, Chairman. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Ήταν πολύ καλό να ακούσουμε αυτούς τους ομιλητές. Γνωρίζω ορισμένους εκ των ομιλητών, όπως τον κύριο Καγό, προηγούμενες ε, συναντήσεις μας. Και Μπορώ, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με όσα είπατε ότι όταν έχουμε αριστεία στην επιστήμη σημαίνει ότι θα έχουμε και αριστεία στην οικονομία για το μέλλον. Αυτό πρέπει να αναφερθεί όταν ε, συζητάμε για το πρόγραμμα έρευνα και νομίζω ότι είναι ένα βασικό μήνυμα που πρέπει να ακούσει το Συμβούλιο και Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές θα ψηφιστεί τελικά το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο μπορεί να πει μόνο ναι ή όχι. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση που έχει να κάνει με τον τελευταίο μιλητή, ο οποίος είπε ότι ε, πρέπει να δώσουμε μία έμφαση στις αναδυόμενα τμήματα και όπου δεν υπάρχει ακόμα η αριστεία. Εγώ προέρχομαι από την Ουγγαρία και ούτε η επιστήμη ούτε η οικονομία λειτουργούν καλά εκεί. Ποια θα ήταν η δική σας πρόταση για αυτές τις χώρες που είναι σε αυτήν την κατάσταση να μην ε, καθυστερούν ε, ίδιες αφενός αλλά να μην καθυστερούν ούτε και εσάς. γιατί το χειρότερο θα ήταν να χαθούν ε, οι δεσμεύσεις, ε, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ε, από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, πώς πρέπει να οικοδομηθούν στρατικές και να δεσμευτεί ο καθένας στα project. Για μένα ως πολιτικός θα ήταν πάρα πολύ ε, δύσκολο ε, να βλέπω ότι θα χάνει η χώρα μου πραγματική χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χέρτσοκ. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους α, ε, α, ανθρώπους που μίλησαν με διαφώτισαν σε πολλά σημεία. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Μαξ Planck γιατί με τα στοιχεία του μας βγάζει από τον μόνιμο ευρωπαϊκό αυτισμό και μας φέρνει σε σύγκριση με το διεθνές περιβάλλον. Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά αν κανείς τα συγκρίνει με ένα παγκόσμιο κλίμα που απεικονίζεται ακριβώς στην κλίση των καμπυλών που δείχνουν την αύξηση των δαπανών στους δύο κύριους ανταγωνιστές στην Κίνα και την Αμερική. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι μόλον ότι προέρχομαι από μικρή χώρα που δεν είναι πολύ εύκολο να το πει κανείς, επιμένω ότι ο μόνος δρόμος για την Ευρώπη είναι η αριστεία σε αυτήν οφείλουμε να επικεντρωθούμε. Και ταυτοχρόνως να καλέσω τον φίλο μου τον κύριο Γιάνν Σμίτς να βρούμε τα μέσα έτσι ώστε οι χώρες που καθυστερούν στη στρατηγική της Λισαβόνας μέσω της συνεργασίας διαρθρωτικών ταμείων και ερευνητικών προγραμμάτων να υποστηριχθούν με άμεσο τρόπο στην ανάπτυξη αριστείας. Η αριστεία είναι μια διαδικασία που δεν επιδέχεται δημοκρατική εξομάλυνση είναι εξαιρετικά αριστοκρατική διαδικασία και πρέπει αυτή να ενισχύσουμε την αριστοκρατία του πνεύματος και συνεπώς την αριστοκρατία της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστούμε για αυτούς τους εξαιρετικούς ε, ομιλητές. Μπορείτε να μας πείτε το πώς είναι δυνατόν οι υποτροφίες να χορηγούνται με συντομότερες διαδικασίες, γιατί ε, έχουμε πει ότι έτσι μπορούμε να έχουμε και αριστεία και σε αυτούς που ζητούν τις υποτροφίες. Επομένω, θα πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσει βέβαια με κάποια χρονική άνεση, αλλά να διεκπληρώνεται η διαδικασία συντομότερο. Και αντίστοιχα είναι αποτελεσματική και η χορήγηση των πληροφοριών, η ενημέρωση της υποτροφίας. Ευχαριστώ. Καρβάλιο. κύριε Καρβούδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους όσους ομίλησαν και για όλα όσα μας πρότειναν και επίσης έχω κάτι να σας ρωτήσω τι γίνεται όσον αφορά την αριστεία, όσον αφορά την πορεία προς την αριστεία, διότι θα πρέπει να χαιρετήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει τα γεωγραφικά κριτήρια ή άλλου είδους προϋποθέσεις από την αναζήτηση των καλύτερων λύσεων και επίσης θα πρέπει έτσι να δούμε ε, πώς θα μπορέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να εντάξουμε την αριστεία στο, στο πρόγραμμα 2020 και ακριβώς εδώ έχουμε για την έννοια αυτής της κλίμακας, της διαδρομής, της σκάλας ε, προς την ε, αριστεία και να λάβουμε υπόψη και τα μικρότερα κέντρα αριστείας, τα μικρότερα κέντρα έρευνας. Και προσοχή όμως, ένα είναι αυτό και άλλο είναι ε, η δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων, το capacity building, ε, γιατί θα πρέπει να ε, συνδυάσουμε το Horizon 2020 με την προσπάθεια για την δημιουργία και εκμετάλλευση δυνατοτήτων και επομένω να βοηθήσουμε και τα μικρότερα ερευνητικά κέντρα, αυτά τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Το Horizon 2020 θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο που να καλύπτει και αυτά τα μικρά ερευνητικά κέντρα ε, ήδη μας, ε, μας είπαν για τέτοιες περιπτώσεις. Παρακαλώ, πέστε μας και άλλα παραδείγματα. Πώς θα κάνουμε την εφαρμογή αυτής της σκάλας προς, το, προς την αριστεία στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020. Η πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κουτιέρες Κορτίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, έχουμε τώρα διάφορα επί των οποίων θα ήθελα να σας ε, μιλήσω. Με προβληματίζει και με προβληματίζει ανέκαθεν το ότι έχουμε πρόβλημα για την ανέβρεση ε, ανθρωπίνων πόρων που να αφιερωθούν στην ε, έρευνα. Το Μαρικυρί δεν επαρκεί, το ξέρουμε όλοι. και είναι λάθος ο διαχωρισμός Κιουρί από το Horizon 2020 όσον αφορά την έρευνα. Να μην έχουμε την έρευνα χωριστά από την κατάρτιση. Και πάνω σε αυτό έχω να σας πω τα εξή. Ε, ο κύριος από το Max Planck. Από ό,τι γνωρίζω στην ε, Γερμανία έχετε project κοινή κατάρτισης και σπουδών κοινών μεταξύ πολλών πανεπιστημίων. Είναι δυνατόν τις υποτροφίες να τις ε, συνδυάσετε κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να συνδυαστεί ο δημόσιος με το ιδιωτικό τομέα. Παρακαλώ ενημερώστε μας και να εντάξουμε την εμπειρία σας στο πρόγραμμα. Τώρα για τα πανεπιστήμια. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση από τον φορέα των ε, πανεπιστημίων. Όμως αυτή η ενδοσκόπηση είναι πληγή. Είναι κάτι το οποίο βλάπτει όλο τον κόσμο και αυτό σας ρωτώ. Μπορείτε να προβείτε σε κάποιο είδους υποχρεωτική αξιολόγηση των ε, πανεπιστημίων. Και να αξιολογηθεί όλη η διαδρομή, όχι μόνο σημειακά. Και αυτό να ισχύει και για την απονομή των υποτροφιών. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μέχρι ένα σημείο νομίζω. Τρίτη ερώτηση. Θα προσφύγει ενδιαφέρον να συνδυάσουν τα διαφορετικά ταμεία στις πιο αδυνατές χώρες με τις χώρες της αριστείας. Και έτσι να υπήρχε κάποιο είδου ε, βοήθεια από πλευράς των πανεπιστημίων αριστείας. Μια τέτοια πρόταση να την ε, προωθήσουμε και έτσι να υπάρχει μεταφορά πόρων, να βοηθηθούν οι πιο αδύνατοι. Και έτσι να υπάρχει βοήθεια από τα διορτικά ταμεία. Ο Μία ερώτηση έχω να κάνω, η οποία ουσιαστικά ετέθηκε για τους συναδέλφους. Αν η αριστεία πρέπει να παραμείνει η βασική αρχή και από αυτού συμφωνούμε, πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα των χωρών εκείνων που πολύ απλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο αυτό στην Επιτροπή μας. Υπάρχει μια απόφαση και μια πρόταση, μια ιδέα για έναν ανταγωνισμό όπου οι χώρες αυτές και οι χώρες που είναι ήδη προηγμένες στο τομέα αυτό θα έχουν μια σύνδεση. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Θα θεωρείτε ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα μια τέτοια πρόταση γιατί αν το θέλουμε αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε ως περιφερειακό σημείο θα πρέπει να το θέσουμε στο επίκεντρο των προσπάθειών μας όχι μόνο να μείνουμε στο επίπεδο του 3% αλλά να δημιουργηθεί και ένα ξεχωριστό αποτελεσματικό εργαλείο. Ευχαριστώ, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις πολύ καλές εισηγήσει όλων των ομιλητών. Θα ήθελα να θίξω δύο σημεία μόνο. Από όλες τις εισηγήσει κατάλαβα το κριτήριο για το πρόγραμμα Horizon 2020 θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός στην αριστεία. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά ας το υπενθυμίζουμε κάθε φορά ότι πραγματικά είναι τεράστια ανάγκη να το θυμόμαστε αυτό. κοιτώντα ε, βάσει των δημοσιεύσεων στον πίνακα που μας παρουσιάσατε, πού βρισκόμαστε, έχουμε ένα, δύο, τρία, μάλλον από 10 πανεπιστήμια σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση ως προς την αριστεία. 9 από τα 10 είναι ε, αμερικάνικα και μόνο το Ίδρυμα Max Planck ε, παρουσιάζεται στον κατάλογο αυτό. Λέμε λοιπόν ότι θέλουμε την αριστεία, αλλά θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε όλα αυτά, γιατί σε παγκόσμιο προσκήνιο θα χάσουμε και συμφωνώ αυτά που είπαν και πολλοί συνάδελφοι και η συνάδελφος Χέρτσοκ ότι αν δεν ε, προσανατολιστούμε στην αριστεία δεν θα υπάρξει αντιμία και από αυτό εξαρτάται και η οικονομία μας και η κοινωνία μας. Ε. Το κριτήριο λοιπόν της αριστείας θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό κριτήριο και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ERC και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Horizon 2020. Αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά όλους είναι όλα τα κράτη-μέλη να υποστηριχθούν στις προσπάθειες που καταβάλουν. Να θέσω μία ερώτηση. Πώς ε, θα καταφέρουμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα αυτό το δρόμο προς την αριστεία. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις γιατί ε, προφανώς ε, είναι έξυπνο να συνδυάζουμε τα μέσα συνοχής με το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά θα ήθελα να ακούσω και άλλες προτάσεις και ένα ακόμα στοιχείο για συγκεντρώσουμε τους πιο ικανούς θα πρέπει να αναφερθούμε και στις γυναίκες και ίσως αυτό δεν το ανέφερετε γιατί ε, είσαστε όλοι άνδρες οι ομιλητές όχι, σας το αναφέρετε αλλά πώς μπορούμε λοιπόν να υποστηρίξουμε και τις γυναίκες στην έρευνα και την ανάπτυξη Ευχαριστούμε κύριος Μπερλίνγκουερ Ευχαριστώ και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τους υπολείπους. Ε, πολύ θετική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας. Δύο θέματα όμως ε, θέλω να θίξω, δύο ερωτήσεις. Ε, η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά στην έρευνα, αλλά χάνει αδέφος στον παγκοσμίο ανταγωνισμό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα εθνικό ίδρυμα επιστημών και το ίδιο και οι Κινέζοι και οι Άπωνες. Εμείς έχουμε 27 Εθνικά Συμβούλια Ερευνάς ε, και έχουμε βέβαια και κάποια εξαιρετικά όπως ε, το Max Planck. Ο ευρωπαϊκό πρόβλημα επίσης είναι το θέμα της ολοκλήρωσης, δηλαδή ε, διάφοροι τομείς. Πρέπει να το δούμε αυτό εις βάθος. Εγώ νομίζω ότι από τότε που υπάρχει το πρόγραμμα πλαίσιο έχουν μεγάλα βήματα προς τα μπρος και σήμερα έχουμε ένα πολύ εύρωστο οικοδόμημα. Όμως πρέπει να εργαστούμε γιατί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, ευρωπαϊκό συντονισμό ε, των ερευνών σήμερα, γιατί πρέπει να ενισχυθεί. Υπάρχει ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, βεβαίω ε, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά είναι βήματα προ τα μπρος, αλλά δείτε πόσο δυσκολευτήκαμε να οθήσουμε τη διαδικασία της Μπολόνια, που τις προάλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όθησε ε, πολύ αποφασιστικά. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να ενισχυθούν όλα αυτά, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα, ε, μία κληρονομιά ερευνητών είναι μία από τις οδούς που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και κάτι τελευταίο, δεν γίνεται μεγάλος λόγος για διαδεδομένη επιστημονική κουλτούρα. Αυτό διαφέρει από την επιστημονική έρευνα. Δηλαδή για επιστημονικά κέντρα για επιστημονική μόρφωση. Πρέπει να υπάρχει ενίσχυση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει μια δράση για να μεγενθηθεί η επιστημονική κουλτούρα της Ευρώπης, γιατί όλα αυτά στη συνέχεια τροφοδοτούν και την έρευνα. Ευχαριστώ, κύριος Τζόνσον. Ευχαριστώ. Θα θέσω την ερώτησή μου στα Σουηδικά. Συμφωνώ απόλυτα με τους προελελήσαντες. Είναι αλήθεια ότι ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Και όπως είπατε και στην αρχή κυρία Πρόεδρε, δεν ε, χρειάζεται να μας πείσετε εμάς ε, για το πόσο σημαντική είναι η έρευνα και η γενοτομία. Ε, θα ήθελα να επανέλθω σε μία ερώτηση ε, στην ε, κυρία Μαντιρέλ. Εγώ προερχόμαι από τη Σουηδία και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προοπτική αριστείας. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως θα πρέπει να εξετάσουμε και την πολιτική πραγματικότητα. Εμείς ε, που εξετάζουμε αυτό το πρόγραμμα από πολιτική σκοπιά, πρέπει να δείξουμε πώς η αριστεία μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη συνεισφορά για το σύνολο της Ευρώπης. Πολλοί συνάδελφοι έθεσαν το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα, γιατί τελικά ε, είναι πολιτική η συζήτηση, η αριστεία, η έρευνα και η καινοτομία. Είναι κάτι που πρέπει να ωφελήσει το σύνολο της Ευρώπης. Ε, έτσι λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η δική σας πρόταση πώς ε, από πολιτική σκοπιά μπορούμε να ενισχύσουμε τη διάσταση της έρευνας, ε, προκειμένου η έρευνα και η καινοτομία να αποτελούν πλεονέκτημα για όλη την Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί αλλά τι μπορούν να κάνουν και οι θεσμικοί φορείς, τα ερευνητικά ιδρύματα κτλ. Το να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των διαφορών ιδρυμάτων είναι κάτι που μπορεί να συνεισφέρει, αλλά θα πρέπει φυσικά να έχουμε κατά νου και τις ε, πολιτικές ε, πραγματικότητες. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, γιατί και η αριστεία ε, προέρχεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά τα ερευνητικά κέντρια κοιτούν και προς την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε την αριστεία στην επιστήμη με την αριστεία στην οικονομία, γιατί αυτό αποτελεί και τη βάση για την καλύτερη μεταφορά know-how στην πράξη. Καλωσορίζω τις ε, πρακτικές της εταιρείας Max Planck και άλλωστε και ο καθηγητής Γκρούς μας παρουσίασε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στην εισήγησή του. Μας είπε ότι κυρίως θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία ακόμα και όταν είναι μικρό το εκάστοτε ίδρυμα. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα για τα άλλα ιδρύματα τα οποία ενδεχομένως να βλέπουν το μέλλον τους σε πιο μεγάλη χρηματοδότηση αλλά να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε με ποιους δείκτες προσμετράται η επιτυχία και πώς δημιουργείται και ένα γενικότερο πλαίσιο για την προώθηση της δημιουργικότητας προκειμένου οι ερευνητές να διευκολύνονται ως προς τη δημιουργική τους διάθεση. Ευχαριστώ, κύριε Αντελκαστήγιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Θεωρώ ότι τόσο υπόθηκαν είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το καθήκον μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Βέβαια, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό. Θέλω να αναφερθώ στην διεθνή διάσταση. Κατά την έποψή μου, ορίζοντα 2020 θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να ανοίξει ο χώρος έρευνα και ενδομίας τη Ευρώπη στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία μονής ε, κατεύθυνσης, ε, δηλαδή να βρούμε πόρους ε, εκτός Ευρώπης, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και την παρουσία των ευρωπαϊκών οντοτυπών σε τρίτες χώρες και να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες με μη ευρωπαϊκές οντότητες σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη βάσει κριτηρίων αμοιβαιότητας. Μάλιστα, εσείς παρουσιάσατε μια σειρά συνεργατικών σχεδίων και κέντρων. Έτσι λοιπόν αναφερθήκατε στο τι συμβαίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δυστυχώς παρά ε, το να ανοίξει αυτό το πρόγραμμα στις τρίτες χώρες ε, χρειάζεται συγκεκριμένο κονδύλι γι' αυτό και δεν αποτελεί αυτό τομέα προτεραιότητα. Όλα εξαρτώνται από αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μία σαφή ε, ανάληψη υποχρέωσης να εκταμιευτούν συγκεκριμένοι πόροι στη διεθνή συνεργασία κατά την άποψή μου θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε ενδυνάμει συμμετέχοντες σε παγκόσμια προγράμματα. Πρέπει να αναφέρω ότι η προτεραιότητα αποτίθεται από το Στρατηγικό Φόρουμ Διεθνή Συνεργασία, αποδυναμώνεται στην πρόταση. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω κάτι που με ανησυχεί οι πολιτικοί περιορισμοί προέρχονται και από προτάσεις ε, όπως η εξής για ένα αριθμό τομέων παρόλα αυτά μία προσέγγιση πιο προσεκτική ίσως ε, θα έπρεπε να ακολουθηθεί για να διαφυλαχθεί το ευρωπαϊκό συμφέρον. Λαμβάνοντας υπόψη μία τέτοια προσέγγιση στην πράξη κάτι τέτοιο μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε δραματικές μειώσεις στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας. Θέλω λοιπόν να τον απτύξετε λίγο περαιτέρω αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτή η διεθνής διάσταση έχει ρόλο να παίξει στον ορίζοντα 2020 και εξακολουθεί να είναι κάπως αδύναμο αυτό το σκέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, μισή ώρα, έτσι έχει η κατάσταση και έχουμε πάρα πολλού που έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο. E Σας παρακαλώ, ένα μισή λεπτό. Συνάδελφος Όκμαρ. Um, uh, Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές. Εμένα μου λείπει μια καθαλική προοπτική σε κάποιες παρουσιάσεις με κάποιες εξαιρέσεις και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια τάση να συζητούμε εδώ πώς ε, θα μοιράσουμε την αριστεία που έχουμε σαν να ήταν αυτό το πρόβλημα αλλά το πρόβλημα είναι η αριστεία που δεν έχουμε έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των παγκόσμιων προοπτικών. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τους προσκεκλημένους μας, μπορείτε να τοποθετηθείτε σχετικά με το πώς η ευρωπαϊκή έρευνα ε, θα μετατραπεί σε παγκόσμια κέντρα αριστεία, πώς θα προσεγγίσουμε περισσότερες διεθνείς προσπάθειες στην Ευρώπη. Ουσιαστικά ακολουθώ την ίδια γραμμή με την κυρία Δελκαστήγιο. Αλλά επίσης πώς θα αντιμετωπίσουμε θέματα όπως να προωθήσουμε την αριστεία σε άλλες περιοχές της Ένωσης μέσω των διαφορετικών ταμείων, γιατί να αρχίσουμε να συζητάμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα πλαίσιο, προκειμένου να βοηθήσουμε όλα τα μέρη της Ευρώπης να αποκτήσουν αριστεία, τελικά δεν θα έχουμε καθόλου αριστεία, γιατί ε, η φιλοσοφία του προγραμμάτου είναι στο ανώτερο επίπεδο να χρησιμοποιηθούν όλε οι προσπάθειε για να κατασταθούμε ακόμη καλύτεροι από όλα μέρη του κόσμου. Θα ήθελα το πάνελ λοιπόν να επανέλθει στην πρόκληση αυτή, πώ θα είμαστε καλύτεροι από του υπολείπου. Για να μην κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για το πώ θα μοιράσουμε κάτι που δεν έχουμε. Ευχαριστώ, Ράνσφορντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να πω ότι από όλες τις παρεμβάσεις που άκουσα σήμερα το πιο ενδιαφέρον μου φάνηκε αυτά που μας είπαν από την εταιρεία Max Planck σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αλλά θα πρέπει να πω ότι όσο πιο πολύ κάθομαι εδώ, τόσο πιο πολύ έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα οργάνωσης των προοπτικών. Δεν σημαίνει αυτό ότι αναφερόμαστε στην ουσία του προβλήματος που είναι η γενικότερη νοτροπία, η γενικότερη διάθεση του σκεπτικισμού, αν θέλετε, για την τεχνολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λείπει λοιπόν αυτό το πρωτοποριακό πνεύμα που, είχα στο παρελθόν, που είχαμε στο παρελθόν και βλέποντας αυτόν τον σκεπτικισμό, συγκρίνοντάς τον με τη διάθεση που επικρατεί στην Κίνα ή σε άλλα τμήματα του κόσμου, πρέπει να πω ότι στην Κίνα ε, υπάρχει μια πείνα για εξυγχρονισμό. Πολλοί κόσμος, ε, χιλιάδες νεαροί αποστέλλονται στην Ευρώπη για να ε, σπουδάσουν την κατασκευή αυτοκινήτων να κοιτάξουν τα αποτελέσματα της τεχνολογίας και της επιστήμης στα ευρωπαϊκά και στα αμερικάνικα κέντρα και επιστρέφουν αυτοί οι νέοι επιστήμονες για να εισάγουν τις κοινωνίες αυτές στα μοντέλα παραγωγής τους. Σας παρακαλώ λοιπόν θα... να κοιτάξουμε πιο πολύ την ουσία του προβλήματος, την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό της κοινωνίας στην τεχνολογία και το να αλλάξει αυτή η διάθεση. Αυτό αποτελεί το πρόβλημα το βασικό. Η χρηματοδότηση μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αποτελεί το βασικό ζήτημα. Και κάτι άλλο. Κοιτάμε το, ιστορικά το πρόβλημα των εφευρέσεων, των ανακαλύψεων και διαπιστώνουμε ότι οι νέες λύσεις οι νέες ανακαλύψεις προέκυψαν πάντα σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Άρα, από ιστορικής άποψης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την θεωρία των μακρών κυμάτων, όπου βλέπουμε ότι επικεντρώθηκαν η πλειονότητα των μεγάλων ανακαλύψεων. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μια προσωμείωση των όρων και των προϋποθέσεων αυτών σε, κανονικούς, ε, σε κανονικές συνθήκες. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο και ένα τον άλλον, ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας κατάστασης μεγάλων αλλαγών. Η εφορία απαιτεί ένα τμήμα των, ε, της κατανάλωσής μας ε, να μην υλοποιείται και πιστεύω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση της επιστημονικής ε, κουλτούρας με την ανθρωπιστική κουλτούρα και πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ποιο είναι το πνεύμα βάσει του οποίου τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στο ζήτημα αυτό και κατόπιν πρέπει να προσέξουμε και το κλίμα που μπορεί να ευνοήσει την ε, καινοτομία, δηλαδή αυτή την ε, παράπλευρη ελεύθερη σκέψη που πιστεύω ότι αποτελεί ενσωματωμένο τμήμα του γενικού κλίματος που πρέπει να δημιουργήσουμε για να γίνουμε μια καινοτόμος περιοχή ως Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Πρόμπη. Πρόντι, με συγχωρείτε, η κυρία Κολάνσκα Μπομπίσκα. Thank ναι, Ευχαριστώ. Συζητάμε εδώ πόσο καθυστερεί η Ευρώπη εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως εγώ ανησυχώ και για τις διαφοροποίησεις που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών στην Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω το διευθυντή του Μαρτς Πλάνκ. Είπατε ότι ανοίγεται νέα κέντρα αριστεία στο Λουξεμβούργο και σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχει τέτοιο κέντρο σε νέο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν θα ήμουν περίεργη και βλέποντας επίσης τα δεδομένα που μας παρουσιάσετε για ε, το πρόγραμμα συνεργασίας με χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ε, ποια είναι τα εμπόδια ε, στη συνεργασία με τις χώρες αυτές για τη διάδοση της γνώσης κτλ. Αναφέρατε ότι ένας τρόπος ε, να γεφυρωθεί το χάσμα θα ήταν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο διαρθρωτικά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία, είπαν κάποιοι. Εγώ δεν νομίζω ότι το οικονομικό είναι το πραγματικό εμπόδιο εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να με ενημερώσετε λίγο περισσότερο όχι για τα οικονομικά εμπόδια της συνεργασίας και της διάδοσης της αριστείας, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριο Στόια. Ε, Κυρία Τόια, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να πω ότι και εγώ θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρουσε τις σημερινές παρεμβάσεις. Να θέσω μια ερώτηση, ίσως ε, κάπως ε, ακαθόδη γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Η κυρία Μαντουρέλ έθεσε κάτι δύσκολο, μια δύσκολη ερώτηση. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε ή να μετρήσουμε την αριστεία. Αν το κριτήριο της αριστείας είναι αυτό που καθορίζει συγκεκριμένα τμήματα του προγραμματός μας, εμείς ε, ως νομοθέτες έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιος αποφασίζει βάσει του κριτηρίου της αριστείας, ε, ε, με ποια κριτήρια εφαρμόζεται αυτό το κριτήριο, υπάρχει στη διαφάνεια. βεβαίω αυτό δεν πρέπει να το αποφασίσουμε εμείς, αλλά έχουμε την ευθύνη να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί οι πόροι, κυρίως αν πρέπει να τους αυξήσουμε προ ορισμένε κατευθύνσει, θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη διαφάνεια και με αντικειμενικότητα. Κάτι που σήμερα είναι δύσκολο για μα για να αξιολογήσουμε. Πώ μπορούμε να το πράξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Τόια να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Γκάγκο για να κάνει μια πρώτη απόπειρα απάντηση. Έχουμε καθυστερήσει κατά μισή ώρα, όπως σας είπα. Δύο λεπτά σας παρακαλώ για τις απαντήσεις. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Γκάγκο, ο καθηγητής Γκάγκο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω εντάχει να διεξέλθω μία-μία τις ερωτήσεις που έθεσαν ε, οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Όσον αφορά αυτήν την κλίμακα, την σκάλα προς την αριστεία, θέλουμε έτσι να προωθήσουμε την αξιόλογη έρευνα στις χώρες. Στις χώρες όπου οι δυνατότητες ε, ακόμα είναι σε χαμηλό επίπεδο. Υπάρχουν όμως ε, αξιόλογα ιδρύματα, αξιόλογοι άνθρωποι. Δεν είναι η καλύτερη ιδέα εντυπωσιακά, θεαματικά κανείς να αντιτίθεται στο πρόγραμμα και να μην, να μην βοηθάει ούτε την συνεργασία ούτε τα, τα διορθωτικά ταμεία γιατί καμία χώρα δεν έχει μπορέσει από μόνη της να κάνει κάτι χωρίς ε, διεθνή συνεργασία. Η διεθνή συνεργασία όσον αφορά έρευνα, τεχνολογία, επιστήμη είναι κάτι το απαραίτητο εκ των νουκάρευ γιατί δεν θα πρέπει επομένω να υπάρχει απομονωτισμός. Δεν είναι δυνατόν επομένως κανείς να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του χωρίς να μπορέσει να ξεκινήσει, να ενισχύσει την δικτύωση με άλλα κέντρα αριστείας σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε τα μέσα πολιτικής που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία του Horizon 2000 ας πούμε, τα μέσα που, μέσω των οποίων απονέμονται βραβεία αριστείας κάθε χρόνο στα κρατημέλη. Αλλά υπάρχουν πολλά, πολλά μέσα. Η κατάρτιση, το άνοιγμα όλων των ε, project συνεργασίας για υποτροφίες πριν ή μετά τη φάση του διδακτορικού ή για το δεκτορικό. Πολλά, πολλά, πολλά μέσα υπάρχουν και μην ξεχνάτε ότι οι εθνικές πολιτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές και δεν μπορεί να βοηθήσει μόνο ο διεθνής παράγων. Και σε επίπεδο εθνικό είναι εδώ να έχουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση, ευκαιρίες να δίνονται εις τους καλύτερους. Να μην προσιλωνόμαστε στα παλιωμοδίτικα σχήματα και έτσι να μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τέσσερα τι να θα σα αναφέρω. Μέσα σε ένα δίλεπτο, αν είναι δυνατόν, γιατί πρώτα πρώτα θέλω να σα αναφέρω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε κανένα ε, είδου ε, αυτομαστίγωση ε, όσον αφορά το τι κάνουμε εδώ πέρα, γιατί είχαμε την επίσκεψη Αμερικανών και πολιτικών και πανεπιστημιακών και εντυπωσιάστηκαν. Εντυπωσιάστηκαν από αυτά τα οποία συζητούμε. Θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πρότυπο, μοντέλο αυτά το οποίο εδώ προσέχουμε. Δεύτερον, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα για, για, για, τουλάχιστον για το δικό μας δίκτυο πανεπιστημίων κανένα πρόβλημα ούτως ώστε να ε, ε, αγκαλιάσουμε αυτά τα οποία ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων, για τη σταδιοδρομία, για την έρευνα. Γιατί φυσικά όντω υπάρχουν πανεπιστήμια παντού που τα, με, τα, με τα οποία συμμεριζόμαστε τις τι προτάσει τη Ένωση και έτσι μπορούμε να έχουμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης και σε σχέση με, με, με, τους, ε, με, με τις προτάσεις Κομισιόν για όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, όσον αφορά αυτήν την τη σκάλα αριστείας, εμείς ως ε, Ένωση Πανεπιστημίων θεωρούμε ότι θα πρέπει η επιστημονική αριστεία να είναι το μόνο κριτήριο όσον αφορά την ε, κατανομή και διανομή των πόρων. ξέρουμε όμως ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα και ότι όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και έτσι να εκμεταλλευόμαστε τι δυνατότητε, τι υποδομέ, του ερευνητέ παντού. Οπότε και εμεί με τη σειρά μα προτιθέμεθα να συνεργαστούμε για τέτοιου είδου δραστηριότητε και εγώ ο ίδιο ε, στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Το ίδιο κάνουμε και έχουμε και αδελφοποίηση με άλλα πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο της Μάλτας για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τώρα επίσης όσον αφορά την αριστεία. Εμείς ως Πανεπιστήμιο μιλούμε για επιστημονική αριστεία και όσον αφορά την ε, μέτρησή της θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι κάνει το ERC. Τι κάνει το, το Συμβούλιο ERC με, με αυτές τις προτάσεις, με τα πάνελς, με τη, τον ε, αυτοέλεγχο ε, εδώ και κάποια χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα και τώρα. Ε, καθηγητά Βελάσκο έχετε το λόγο. Ο κύριος Γκρίσου παίρνει κατά λάθος το λόγο. Α, συμπαθάτε με λέει. Όχι, παρακαλώ, λέει ο κ. Βελάσκο. Έχουμε ένα σωρό ερωτήσει, οπότε πού να βρούμε το χρόνο για να πιέσουμε. Οπότε και εγώ θα επικεντρωθώ εις δύο σημεία τα πρώτα για, τα, ε, για την επιστημονική αριστεία και στα δικά μα ε, ιδρύματα. Ναι, προσπαθούμε αυτό να κάνουμε, προσπαθούμε να έχουμε τη μεταλαμπάδευση των αποτελεσμάτων τη έρευνα, αλλά θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι ο, ο, και ο Bill Gates και ο Steve Jobs ε, ε, ήταν καινοτόμε επιχειρήσει του, αλλά αυτό δεν ήταν επιστημονική αριστεία. Έχουν όμω τη διάθεσή του επιστημονική αριστεία. Οπότε και εμεί στην Ισπανία ε, προσπαθούμε να. Και, και εμεί στην Ισπανία έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μα και, και πολύ κόσμο βοηθάει. Όμω αυτό δεν είναι άριστη καινοτομία. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι του πόλου τη αριστεία, ε, τι χώρε οι οποίε προσπαθούν να, να, να, τα καταφέρουν. Τι να σα πω, ποια είναι η λύση, δεν ξέρω. Ε, Ακριβώ η μεταλαμπάδευση τη γνώση είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει όντω να είμαστε φάνταστοι και να βρίσκουμε τι λύσει. Και οπότε. Ρώτησε κάποιο, κύριε Νίμπλε, ποιο ήταν. Ε, τη συμμετοχή των γυναικών. Το Συμβούλιο Έρευνα, το ERC, Πρόκειται για μια διαδικασία που συνεχώς επιδέχεται βελτιώσεις και διορθώσεις και προσαρμογές. Έχουμε διαδρομή δεκαετία. Στη ΔΕ, Γερμανία, έγινε μελέτη σχεδόν το ρόλο των γυναικών, των γυναικών αφού κάνουν παιδιά Επίσης ε, αντίστοιχα ισχύουν και για τους άντρες όταν πηγαίνουν στο στρατό. Άρα και αυτό έχει σημασία, παράγοντας που έχει σημασία για την επιτεύξη της αριστείας. Γκρούς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν θέλει κανείς να κάνει την Ευρώπη ανταγωνιστική, θα πρέπει να ενισχύσει τους λιγότερο ισχυρούς και να κάνει ισχυρότερους τους ήδη και γι' αυτό και σας παραπέμπω στην ενοποίηση της Γερμανίας. Ο φορέας Max Planck έχει μονάδες ευέλικτες. Χάρη σε αυτές έχουμε συγκροτήσει ιδρύματα. Και τα ιδρύματά μας στην Δυτική Γερμανία είναι το ίδιο αξιόλογα με τα ιδρύματα στην Ανατολική Γερμανία. Άρα δουλεύουμε σε όλα τα επίπεδα και με πολλά πλαίσια. Η επένδυση στους επιστήμονες θα πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε σχολές έρευνας. Έχουμε στενή συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια. Μιλούμε και για το τι θα γίνει με χώρες που δεν είναι και τόσο πρωτοπόρες από πλευρά επιστημονικής και έχουμε επομένω. και κάποια και, και, χρηματοδότηση που την κάνουμε σε ξένες χώρες. Έχουμε προγράμματα που τα τρέχουμε σε άλλες χώρες όπως την Πολωνία. Τα λέμε μοντέλα ακολουθίας και έχουμε συνεργασία με αντίστοιχου πολωνικούς φορείς και έτσι περνάει η χρηματοδότηση εκεί πέρα. Οπότε για να εκμεταλλευτεί, για να δημιουργήσει κανεί νέε δυνατότητες θα πρέπει να βρει φρέσκα μυαλά αλλά και αφού τα βρει να τα εντάξει στο σωστό πλαίσιο. Να, τα διευθυντικά ταμεία, να, το Ταμείο Συνοχής πώς μπορεί να βοηθήσει για να έχουμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Όμως χρηματοδότηση κάποιου προγράμματο, είτε πρόκειται για το ERC, για το Marie Curie, όποιον είναι απαιτείται ούτω ώστε κανείς να έχει κάτι θεσμικού χαρακτήρα μιλάμε για διαδρομή πενταετή έως δεκαετή και κατόπιν η κάθε χώρα φυσικά μετά παίρνει τη σκητάλη και συνεχίζει αφού δεν δοθεί η αρχή όθηση. Πού να προφτάσω να σας πω αυτά που θα ήθελα. Ήδη, ήδη υπερεύει το όριο. Ευχαριστούμε τους κυρίους καθηγητές που σεβάστηκαν το χρόνο και θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαντουρέλ για να κλείσει αυτό το πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, θα χρονοτριβήσω πάνω από ένα λεπτό γιατί οι βουλευτές ήρθαμε εδώ σήμερα να ακούσουμε εσά. Ε, εγώ απλώς ε, θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους ομιλητές και όλους εσάς που θέσατε ερωτήσεις και κάνατε σχόλια. Μπορώ να πω ότι σημείωσα όλες τις προτάσεις σας, όλα όσα κρίνετε θετικά και όλα όσα θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξουν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν ε, θα κάνω πολλά σχόλια, αλλά θα επικεντρωθώ σε δύο σημεία. Το θέμα της αριστείας ε, που επανειλημμένα αναφέρθηκε στη συζήτηση. Η συγκητρία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι θα πρέπει να ανταγωνιστούμε βάσει της αριστείας, αλλά ούτε έχω καμία αμφιβολία ότι πρέπει να διευρύνουμε τον αριθμό των ε, άριστων ερευνητών. Και αυτό δεν αρκεί με τα διορθωτικά ταμεία. Πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα επί των οποίων συζητάμε και μάλιστα πρέπει να δούμε και το θέμα της κατάρτισης. Ε, ήδη έχουμε πάρα πολλές ιδέες κατά νου. Και ένα τελευταίο θέμα για τον προπολογισμό. Αναφέρθηκε γι' αυτό κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τι δράσει Marie χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να σα πω ότι υπάρχει συμφωνία σε όλε τι ομάδε στο να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα για το σύνολο του Οριζόντα 2020, γιατί πιστεύουμε ότι δεν αρκεί ε, αν ε, λάβουμε υπόψη ότι στο ίδιο πρόγραμμα έχουμε έρευνα και καινοτομία για πρώτη φορά. Το επίπεδο επιτυχίας που θα έχουμε θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες, αλλά θα το υπερασπίσουμε αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε καλά μέσα για να προσεγγίσουμε και ιδιωτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, ίσως δεν το συζητήσαμε τόσο σήμερα, αλλά πιστεύω ότι θα ανακύψει και στα επόμενα πάνελ. Αυτά από μένα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαιρετική σας συνεισφορά για να αποτελέσει επιτυχία το πρόγραμμα αυτό. Επιτυχία πολύ επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, να αλλάξουν ε, τώρα συμμετέχοντες ε, στο πάνελ και ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες στο πάνελ αυτό.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 Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ. Καθίστε. Ο κύριος Λάμπερτς ήρθε. Ε, Να ξεκινήσουμε τις εργασίες, ε, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε. Abbiamo tre quarti d'ora di ritardo qui. Κατά 45 λεπτά. Λοιπόν, πρέπει να αναθεωρήσουμε τους χρόνους. Θα ήθελα σας παρακαλώ να καθίσετε ή να βγείτε. Dobbiamo cominciare. Πρέπει να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Οι εργασίες αυτού του πάνελ ε, θα παρουσιαστούν από τον συνάδελφο Ματίας ε, για 5 λεπτά και κατόπιν 10 λεπτά θα έχουν στη διάθεσή τους οι ομιλητές αντί για 15. Σας ευχαριστώ όλους γιατί ε, όλοι ενημερωθήκατε και δεκτήκατε να προσαρμοστείτε σε αυτή τη μείωση του χρόνου. Έτσι λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ματίας. Ε, σας ζητώ συγγνώμη για το θόρυβο στην αίθουσα, αλλά ε, πιστεύω ότι μόνο αν αρχίσουμε τις εργασίες ε, μπορούν όσοι θέλουν να συζητήσουν να περάσουν έξω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι όλοι όσοι περιβρίσκονται στην αίθουσα αυτή γνωρίζουν γιατί βρισκόμαστε δει και εδώ και ποιο θέμα συζητούμε. Εγώ δεν θα μιλήσω πέντε λεπτά, πολύ λιγότερο, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι το σημαντικό είναι να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους εδώ, ε, που ήρθαν να συζητήσουμε τις μεγάλες αυτές ε, κοινωνικές προκλήσεις και στην περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάμε, θα κάνω μια μικρή απερίθμηση. Αλλά ε, μόνο για την περίπτωση την απίθανη που κάποιο δεν γνωρίζει γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη και τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα μέσα από αυτό το πρόγραμμα ορίζοντα 2020. Έχουμε έξι εκθέσεις ε, και δύο ε, εκθέσεις για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας μαζί με τον συνάδελφο Λάμπερτ. Αυτές είναι μεγάλες προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και ενώπιον αυτών έχουμε στη διάθεσή μας ένα σύνολο μέσων και δυνατοτήτων για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση όπου παρουσίασε έξι επιλογές, μία εξ αυτών υγεία και οι δημογραφικές αλλαγές και ευημερία, το το δεύτερο είχε να κάνει με, τη διατροφική ασφάλεια, με την επιστηστική ασφάλεια και με την αηφορία των γεωργικών, των θαλάσσιων πόρων και εγώ θα ανέφερα και την βιολογική οικονομία. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια αποτελεσματική, πιο καθαρή ενέργεια. Τέταρτη πρόκληση έχει να κάνει με τις μεταφορές που ε, πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και πράσινες. Ε, το τέταρτο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, με τις πρώτες ύλε και την αποδοτικότητα των πόρων και η έκτη πρόκληση έχει να κάνει με ε, πιο καινοτόμε και πιο ασφαλείς και συμμετοχικές κοινωνίες. Αυτές είναι επιλογές που έχουμε επιτάπητος και επ' αυτών εμείς προσκαλέσαμε ε, εδώ τους ομιλητές για να μας πούν αν πρόκειται για σωστές επιλογές και να δούμε σε ποιο βαθμό πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά δεν θέλω να χάνουμε περισσότερο χρόνο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ναι, οριζόντια. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, πρέπει να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα και πρέπει να δούμε πού θα επικεντρώσουμε την απάντησή μας. Ε, όμως, όπως ξέρετε, αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται μέσα σε 7 χρόνια. Εμείς συζητούμε τώρα ένα πρόγραμμα για 7 χρόνια και γι' αυτό πρέπει να έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να διαρθρώσουμε τις αλλαγές και τις ε, ουσιαστικές και να δώσουμε μια βιώσιμη απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε. Και αυτή είναι η έβδομη πρόκληση, θα έλεγα εγώ, του ορίζοντα 2020, δηλαδή πώ θα υπάρχουν εγγύσει και προϋποθέσεις ε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να μην είναι αυτό το πρόγραμμα ένα πρόγραμμα μόνο 7 χρόνων, αλλά να το καταστήσουμε ένα πρόγραμμα αλλαγή των κοινωνιών και ιδίω τη Ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ματίας. σα ευχαριστώ που ήσασταν και σύντομοι. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάτου, που προέρχεται από ε, το Τμήμα ιατρική. Uh, Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Χαίρομαι που σα μιλώ σήμερα. Όπω ακούσατε, μα ζήτησα να περιορίσουμε τι παρουσιάσει μα σε 10 λεπτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να καταφέρω να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, λοιπόν, σε 10 λεπτά σε ό,τι αφορά την παγκόσμια υγεία ως ε, πρόκληση της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, προκλήσεις για τις ε, λοιμώτες ασθένειες, που αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια βασική πρόκληση είναι να βρεθούν εργαλεία για να καταπολεμηθούν οι ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλες υπήρους οι μεταδοτικές ασθένειες και μη μεταδοτικές ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα και η αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων προαπαιτεί τη συνεργασία μεταξύ πολλών ε, παραγόντων και είναι βασικό λοιπόν να τονωθούν και να επιταχυνθούν αυτές οι εξελίξεις γιατί αυτές οι προκλήσεις δεν απειλούν μόνο τη ζωή των άμεσα εμπλεκόμενων αλλά και υπονομεύουν την εθνική και παγκόσμια οικονομία. Πρόκειται για κάτι που αφορά και το ιστορικό και το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελενοσία, η φυματίωση και το AIDS από, μόνο του, από μόνα τους κάθε χρόνο κοστίζουν τη ζωή σε 4 εκατομμύρια κόσμος και άλλες παραμελημένες ασθένειες που βλέπετε, κοιτώντας το ποσοστό θνησιμότητα για διάφορες λοιμώδεις ασθένειες. Και επίση ε, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε και σε ό,τι αφορά την σχετική αναπηρία που προκύπτει από ασθένειε. Αντίθετα με αυτά που περιμένει κανεί, ίσω κάποιοι από αυτού ε, του ασθενεί αποτελούν σημαντική ε, απειλή για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω για παράδειγμα στην περίπτωση του AIDS και τη φυματίωση. Πάνω από 2,3 εκατομμύρια κόσμος ζει με το HIV στην ευρωπαϊκή περιφέρεια μέχρι το τέλος του 2010. Πρόκειται για μια επιδημία. Και αυτό, σε αυτό προστίθονται και τα περιστατικά και τα συμπτώματα θυματίωσης σε άτομα με HIV. Έχουμε 49 α, νέες μολύνσεις και 7 θανάτους κάθε ώρα από φυματίωση στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια. Να αποτελεί λοιπόν η φυματίωση μια πάρα πολύ σαφή και μεγάλη ε, πρόκληση για την παγκόσμια υγεία και για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαϊκές ε, ε, κοινωνίες θα ωφεληθούν από οποιαδήποτε πρόοδο της έρευνας και σε βάση της γνώσης αλλά και σε βάση οικονομική. Η υγεία είναι πλούτος. Η επένδυση στην υγεία του πληθυσμού αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης και του ανταγωνισμού. Όπως ε, όσο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα χρειάζεται να εργάζονται όλο και πιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι υγιείς και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο σύνολό της. Αυτό τι σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πιο φθηνούς τρόπους για την παραγωγή ε, με φαρμάκων και εμβολίων. Για παράδειγμα, νέα εργαλεία για την παγκοσμία υγεία. Η βελτίωση της υγείας για τους Ευρωπαίους θα έχει θετικό αντίκτυπο και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά και στα συστήματα κλινικής ασφάλισης. Εκτιμάται ότι, το λιγότερο, ότι λιγότερο από 10% της ε, έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της υγείας δαπανάτε σε ασθένειες, νόσους που επηρεάζουν 90% του κόσμου σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ε, εν τη σωστών ε, μέτρων για την παροχή κινήτρων, δεν ε, γίνεται η ανάλογη επένδυση σε τομείς υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισορροπία προκειμένου να αποδείξουμε τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτά τα προϊόντα της δημόσιας υγείας. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκό επίπεδο στην παγκόσμια υγεία είναι απαραίτητη στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου, ε, του 7ου προγράμματος πλαισίου. Έχουμε 6,1 δισεκατομμύρια ε, συνολική συνδρομή στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη στην υγεία, αλλά μόνο 4% αφιερώθηκε στις ε, βασικές ασθένειες που είναι το HIV, η φυματίωση και η ελονοσία. Και εδώ βλέπετε ένα χάρτη για τον αριθμό των γιατρών που απασχολούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενέκρινε μια ανακοίνωση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παγκόσμια Υγεία το 2010 που υποστηρίζεται από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τα δύο τονίζουν τη σημασία και την ανάγκη συντονισμού καλύτερου ε, σε ό,τι αφορά την έρευνα για την παγκόσμια υγεία και για να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό που επικρατεί στον τομέα αυτό και να τεθούν προτεραιότητες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει συνοχή μεταξύ των προηγούμενων πλαισίων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξωτερικών ε, πολιτικών σε ό,τι αφορά την σχετική πολιτική και έρευνα. Η Ευρώπη έχει εξαιρετικά ερευνητικά κέντρα στον τομέα αυτό. Η ευθύνη για την εξέβρεση λύσεων σε αυτά τα παγκόσμια προβλήματα της υγείας ε, είναι στα χέρια και του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και συνεργασία με τις χώρες που πλήττονται από τις ασθένειες αυτές είναι απαραίτητη προκειμένου να οριστούν οι προτεραιότητες και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην κοινοτομία. Βλέπετε ένα διάγραμμα που δείχνει τον κύκλο της ανάπτυξης και τονίζει ότι χρειάζονται πολλαπλή φορείς από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και φορείς όπως ε, ε, συνεργασίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, θα πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία προκειμένου να υπάρχουν και τα κίνητρα αλλά και η ζήτηση από πλευρά της βιομηχανίας και αυτό μπορεί να το πετύχουμε μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει κίνητρα διατομεακά. Χρειάζονται χρηματοδότηση για την σωστή διαχείριση και σύνδεση της βασικής έρευνη των κλινικών δοκιμών, της εισαγωγής και εφαρμογής των προϊόντων υγείας σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτό θα πρέπει να διατίθεται σε θεσμούς, σε θεσμικά όργανα και οργανισμούς που μπορούν να απευθυνθούν σε όλο τον κύκλο της καινοτομία. Η χρηματοδότηση μηχανισμών θα πρέπει να προσαρμοστεί σε προϊόντα τα οποία μεταβάλλονται ταχύτατα. Και αυτό χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται όχι μόνο μικρές επιδοτήσεις, αλλά και μακροπρόθεσμες, ευέλικτες ε, χρηματοδοτήσεις, όχι βάσει έργων, προκειμένου όλα αυτά να τοποθετηθούν στη σωστή θέση. Οι εταιρικέ σχέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο γιατί συνενώνουν διάφορους εταίρους σε μια νέα εταιρική σχέση που τους επιτρέπει να λαμβάνουν καλύτερους, μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς που ενδεχομένως να ήταν διδεθειμένοι να πάρουν ή μεμονωμένοι βιομηχανικοί φορείς. Τα τελευταία δεκαετία αυτές οι εταιρικέ σχέσεις έχουν αναπτύξει 12 τέτοια προϊόντα για την υγεία και διαθέτουν παραπάνω από 150 προϊόντα σήμερα στην αγορά. Τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα Horizon 2020 για να καλύψει τα, κενή, τα κενά αυτά. Θα πρέπει να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα αυτό για πιο κοινοτομικές μορφές συνεργασίας συνενώντας όλους τους φορείς που χρειάζονται για την ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων. Θα πρέπει να ενθαρρύνουν την καλύτερη έρευνα στα καλύτερα κέντρα, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση. Χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα βάση φακέλου να εντοπίζονται οι καλύτεροι και πιο ικανοί υποψήφοι σε ό,τι αφορά τις κλινικές δοκιμές ε, και σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να απλοποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας προκειμένου να ισχύσουν σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη γιατί αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα α, λύσει συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στην ε, έρευνα έχουν από το αντίκτυπο. Είμαστε κοντά στη δημιουργία εμβολίων για την ενανοσία και σε 50 χρόνια θα έχουμε νέα φάρμακα γιατί μάλλον είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της έρευνας για νέα φάρμακα για την θυματίωση εδώ και 50 χρόνια. Είναι σημαντικό και στον τομέα του HIV να συνεχίσουμε τις, ε, την πρόοδο αυτή για να κινηθούμε ταχαίως προς το μέλλον. Επίσης, ε, η εταιρική σχέση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ε, κλινικών δοκιμών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο. Συμπερασματικά, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος φορέας και χρηματοδότης μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη για την υγεία. Γιατί τα θέματα αυτά όχι μόνο απειλούν τις ζωές των ανθρώπων, αλλά υπονομεύουν και την οικονομική ανάπτυξη και την ε, εθνική σταθερότητα τα νέα προϊόντα μπορούν να μειώσουν το φόρτο που συνεπάγεται μια ασθένεια, το οποίο μακροπρόθεσμα θα απαλλάξει τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς και θα ωφελήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να ανταποκριθούμε στις ε, δεσμεύσεις αυτές, όχι παρά την οικονομική κρίση, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης η επένδυση στην παγκόσμια υγεία θα μας ε, αποφέρει απτά αποτελέσματα προς το συμφέρον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας έκανα να βιαστείτε, αλλά μας ε, έχει φύγει ο χρόνος. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, ε, κυρία Κλάουντια Νεουμπάερ από το Ίδρυμα Σιάνς Σιτουαγιάν. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ευχαριστώ την ε, Ήτρε που ενδιαφέρθηκε να ακούσει την φωνή της κοινωνίας των πολιτών για το ορίζον 2020. Εγώ για πρώτη μου φορά έρχομαι να συμμετάσχω σε μια συνάντηση για σε μια κρόαση για αυτή. Έχω εντυπωσιαστεί και νομίζω ότι τώρα αυτό το που θα πρέπει να κάνουμε είναι το πώς να καταφέρω στα 10 λεπτά να χωρέσω όλα αυτά τα οποία έχω σχεδιάσει να σας πω για περισσότερη ώρα και είμαστε ένα think tank, ένα think tank μη κυβερνητική οργάνωση. Ε, και το θέμα μας είναι τι είδου επιστήμη χρειάζεται η κοινωνία. Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι. Είναι το να εκμεταλλευτούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητε για κοινωνία των πολιτών και για την, για, για την, για την επιστήμη, ούτως ώστε έτσι, να προωθηθεί η συνεργασία των επιστημών για να υπάρχουν επομένω πολλέ εναλλακτικέ και επιλογέ. Ήδη επομένω εμεί έχουμε ε, προσπαθήσει να αναζητήσουμε ε, το στρατηγικό πλαίσιο. Έχουμε το δεδομένη την πράσινη βίβλα του Φεβρουαρίου της Κομισιόν και έτσι είχαμε κάποιο είδους ε, άτυπη συνεννόηση και προγραμματιζόμαστε με την πρώτη αυτή πρόταση της Κομισιόν διότι θεωρούμε ότι έχει συγκεκριμένες απόψεις για ανταγωνιστικότητα, για τη διαχείριση, για τη διακυβέρνηση της επιστημονικής έρευνας. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτά τα που λέει η Κομισιόν αντιστοιχούν ε, ε, σε αυτά τα οποία απαιτούνται. Οπότε θα πρέπει να γίνει κάποιο είδου στροφή στην καινοτομία για, το Horizon 2020. Ε, συντάξαμε μια, μια επιστολή, το στείλαμε στον κύριο Μπαρόσο, αλλά και στο Κοινοβούλιο, εάν θυμάστε, και κατά αυτόν τον τρόπο ε, θα σας αναπτύξω τρεις βασικούς άξονες. Πρώτα-πρώτα για τις ε, προκλήσεις της κοινωνίας. Έχουμε και δύο θεματικά παραδείγματα και την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια σύντομη ε, σημασιολογική ανάλυση εδώ και μπορείτε να δείτε ότι έχουν πάρα πολλούς ε, όρους που έχουν να κάνουν με την αγορά, την βιομηχανία, τη ε, ΜΜΕ και όχι που σχετίζονται με αυτά και όχι με την κοινωνία των πολιτών. Οπότε μπορείτε εδώ πέρα να δείτε τι γίνεται όσον αφορά την πρωτοπορία η πρωτοπορία στην βιομηχανία εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες, αλλά εδώ δεν λέει τίποτα για την κοινωνία των πολιτών ή για τους πολίτες. Οπότε, έτσι κανείς προβληματίζεται. Α, μισό, μισό λεπτό, μισό το λέω η Ορμέλια. Να, τι δηλώνουν οι λέξεις και οι συγχρονίες που χρησιμοποιούνται. Ίσως έχει σημασία. Οπότε, για να δούμε τώρα την σημασία αυτών των λέξεων. Ε, όταν μιλούμε για βιωσιμότητα, τότε βέβαια υπάρχει μια διαφορά μεταξύ βιώσιμης έρευνας και βιώσιμου περιβάλλοντος και βιώσιμων υποδομών. Και όταν μιλούμε για πολίτες, ε, το θέμα είναι αν κανείς τους θεωρεί παράγοντα παθητικό ή ενεργητικό δημιουργικό. Οπότε, οι προκλήσεις για την κοινωνία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία και όχι τόσο για το δεν έχουμε τόσο σχέση με τους πολίτες. Τίποτα δεν αναφέρεται επομένω για την κοινωνία και τους πολίτες. Ε, όμως εδώ καλούνται να παίξουν το ρόλο τους ως καταναλωτές. Όμως οι προκλήσεις για την κοινωνία αφορούν κάποια δίκαιη συμμετοχή και μια που μιλούμε για την αριστεία έχουμε βεβαίως την βιομηχανία που σχετίζεται, αλλά εδώ δεν αναφέρεται από την κοινότητα των πολιτών. Δεύτερον, έχουμε δύο παραδείγματα. Πρώτα πρώτα για τη γεωργία. Είναι δύσκολο όπως είναι τώρα τα πράγματα να καταλάβουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως σας υπενθυμίζω ότι εάν δείτε τι προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί FP3, βλέπετε εκεί μέχρι FP6 μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι αρκετά τα χρήματα καταρχήν. Όμω, αν κανεί κοιτάξει πιο προσεκτικά για την βιολογική γεωργία και την έρευνα, τι ε, χρήματα δίνονται σε σχέση με τη γενική προκοδότηση των προγραμμάτων πλασίων, τότε θα καταλάβετε ότι στην τελευταία, τελευταία στήλη εκεί, ότι δεν υπάρχει καμία αύξηση μεταξύ FP3 μέχρι το FP6 όσον αφορά τα χρήματα που δίνονται για βοήθεια της βιολογικής γεωργίας. Επίσης, εδώ μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση για την χρηματοδότηση, μπορείτε να δείτε τι γίνεται στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, τι, γίνεται με τη βιοτεχνολογία, για τη σχετική έρευνα στη Γεωργία και μπορείτε εδώ να δείτε ότι έχουμε τριπλάσια ενίσχυση της βιοτεχνολογικής γεωργίας. Άρα το θέμα είναι τι θα γίνει με το Horizon 2020 ε, τι, τι κομμάτι του, του προπολισμού θα αφιερωθεί σε κάθε κατηγορία γεωργίας ή, ε, τώρα γιατί από, την, από τον τομέα της ενέργειας το άλλο παράδειγμα μπορείτε να δείτε από τη διαφάνεια ότι μέχρι το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο είχαμε σημαντικούς πόρους του προπολογισμού που γίνανε στην ε, Euratom σε σχέση με το τι προβλέπετε για το πλαίσιο, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως ε, κατέβηκε η χρηματοδότηση στο 30%. 30% από όσα παίρνει η Euratom. Όμως τώρα έχουμε για το Horizon 2020 καλά μαντάτα. Μια που ο προϋπολογισμός εδώ ε, ενισχύει σημαντικά αυτό το τομέα. Όμως Άνοιξε μια ματιά στο τι γίνεται με την αποτελεσματική χρήση ενέργεια, τι γίνεται με την ηλιακή ενέργεια, τι γίνεται με την κατακράτηση και αποθήκευση του άνθρακα το τότε βλέπουμε ότι αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ διφορούμενα, πάρα πολύ πίμαχα και δυσκολεύεται κανείς να ε, καταλήξει στο πώς θα γίνει η κατανομή των πόρων του προπολογισμού μεταξύ αυτών των διαφορετικών κατηγοριών. Τώρα, συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών είναι ο μέγας απόν από το πρόγραμμα. Η επιστήμη στην ε, κοινωνία εξαφανίζεται όμως είναι πάρα πάρα πολύ αυτά τα οποία προβλέπονται σχετικά και αυτό μας εκπλήσει πολύ διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε την συμμετοχική έρευνα την τελευταία 12 ετία με το πρόγραμμα ε, πλαισίο 6 και το 7 Οπότε έτσι έχουμε την κινητοποίηση για την αμοιβαία εκμάθηση ε, και με το, καινούριο πλαίσιο χρηματοδότησης έχουμε ε, ως επιλέξιμες σημαντικές συγκεκριμένες ομάδες και αυτά τα προγράμματα είναι πρωτοπόρα. Όμως τι έμεινε από αυτό. Πάρα πολύ λίγο αν κάνει δει τι ε, συμμετοχικέ προκλήσεις, γιατί θα έπρεπε να είναι πιο εγκάρσια η συμμετοχή και η πρόβλεψη για την ε, κοινωνία. Μόνο σε δύο σημεία αναφέρεται. Για το κλίμα, για τη, εκεί που λέει επίση για την. Ε, για τη συμμετοχική, για τη συμμετοχική κοινωνία αναφέρεται κάτι. Όμως θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, βελτίωση Τη παιδεία όσον αφορά την επιστήμη και επομένως διαπιστώνουμε ότι έχουμε πάρα πολύ παραδοσιακή αντίληψη για το τι είναι η επιστήμη. Ότι ο κόσμος θα πρέπει να μάθει από την επιστήμη αλλά η επιστήμη δεν έχει τίποτα να διδαχθεί από τους επιστήμονες και από την κοινωνία των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, όλες μας οι εμπειρίες από τη συμμετοχική έρευνα αφορούν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον και επομένω. Βλέπετε τι γίνεται όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση πρόκειται για κάτι το οποίο ήδη λειτουργεί και θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς και βοηθάει στην πρόοδο. Όλα ένα και περισσότερο οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών διατυπώνουν ε, τις ανάγκες τους και γίνονται οι πελάτες ούτως είπε, είναι αποδέκτες της έρευνας. Υγεία, περιβάλλον, γεωργία, ενέργεια, μεταφορές, ε, κοινωνική πολιτική, όλα αυτά αφορούν την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και επομένως κάπου ε, εκεί στον, στον, πραγματικό κόσμο υπάρχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστημονική γνώση αντιστοιχεί σε αυτό το οποίο θέλει η κοινωνία. Επομένως, δημιουργούνται κάποιες ε, συμμαχίες μεταξύ ερευνητών και της κοινωνίας. Υπάρχουν κάποια δίκτυα, υπάρχουν ε, διάφοροι φορείς, νομικά πρόσωπα, όπου δημιουργείται μια κουλτούρα, μια εμπειρία συμμετοχής. Αυτό είναι πολύ καλό για την επιστήμη, διότι καθ' τον τρόπο θα έχουμε μια εναλλακτική τεχνολογία, νέες ε, διευθύνσεις, η, σκεφτείτε την οικοτοξικολογία. Ε, αν δεν υπήρχε βοήθεια, πίεση απ' έξω, τότε όλη η πρόοδος θα είχε καθυστερήσει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά προκλήσεων. Ε, δεν θα πρέπει να παίρνουμε αυτονόητα κάποια πράγματα όπως, την, όπως η καινοτομία, η πρόοδος και οι αξίες οι οποίες είναι τα θεμέλια της ε, ανάπτυξης. Μεγάλη διαφορά κάνει η κοινωνία των πολιτών εάν συμπεριληφθεί σε αυτές τις εξελίξεις. Ακριβώς ε, όσο σημαντική είναι και η βιομηχανία. Βεβαίω και οι προτάσεις της ε, Ήτρες, την πρώτη έκθεση για την συμμετοχή της των πολιτών τις εγκρίνουμε και να οι κανόνες για τη συμμετοχή και ο κανονισμός ε, επίσης ε, στο άρθρο 12 και 13 προβλέπει σχετικά και όλα αυτά αφορούν την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαριστούν περισσότερο και να λάβουν υπόψη στους κανόνες συμμετοχής τι λέει το σημείο 10, τι θα πει ε, νομικό πρόσωπο λέει εκεί σε σχέση με την κοινή των πολιτών αλλά εδώ δυστυχώς ο χρόνος μου τελείωσε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να καθησυχάζω όλους ε, τους ομιλητές ότι πέρα από το ότι σας ακούμε, διαβάζουμε ε, και όσα κείμενα μας αφήνεται και τα Τώρα η κυρία Μικελώνα, η οποία είναι αντιπρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης για τη Βιολογική Οργία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ και την ε, Κλάουντια που διευκόλυνε το έργο μου γιατί είπε πάρα πολλά στοιχεία για την ε, γεωργική έρευνα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αναφερθώ στα κύρια σημεία της παρουσίασής μου. Όπως σας είπα, είμαι αντιπρόεδρος της Νόσης για τη Βιολογική Γεωργία, αλλά εδώ εκπροσωπώ την τεχνολογική πλατφόρμα για την βιολογική γεωργία και έρευνα. Θα μιλήσω αγγλικά και θα προσπαθήσω να μην επικεντρωθώ τόσο στην Ιταλία, αλλά θα επικεντρωθώ σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πολύ σύντομα, ποιες αλλαγές ε, τροφοδοτική γεωργία και πώς μπορεί να συνεισφέρει η γεωργία σε μια μερική λύση. Προσπαθώ να αναφέρω τα κυρία και νομίζω ότι η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων μας είναι η κύρια κοινωνική αλλαγή πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η γεωργία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ακόμη και αν η γεωργία είναι με ψηφία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αγροτικές περιοχές, ακόμη και αν μεγαλώνουν όσο περισσότερες οι πόλεις. Οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να δουν, ζουν στην επαρχία. Έτσι λοιπόν ό,τι συμβαίνει δεν ε, έχει επιπτώσει μόνο στους γεωργούς αλλά και στους κατοίκους αλλά και φυσικά σε όσους τρώνε αυτά που παράγει η γεωργία. Έτσι λοιπόν ε, το μέλλον της ε, γεωργίας επηρεάζει όχι μόνο τους γεωργούς αλλά το σύνολο του πληθυσμού και όλους τους πολίτες. Ε, και όχι μόνο στους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι μετά την υποβάθμιση του συστήματος στη δεύτερη ε, πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή όπου η Γεωργία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και κατόπιν έχουμε την επιστημιστική ασφάλεια ανασφάλεια ανάλογα πώς το βλέπει κανείς αλλά επίσης και τους ελλειπείς πόρους και την έλλειψη κοινωνικής συνοχής και τέλος την υποβάθμιση του εδάφους και πρέπει να τη μετατρέψουμε σε προστασία του εδάφους. Εμείς ε, εκπονούμε τουλάχιστον τρία κυρία γράφα που μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Δεν ε, θα αναφερθώ περαιτέρω, αλλά αποτελούν το όραμα για τη Γεωργία τα γράφα αυτά. Ε, είναι η ατζέντα για την έρευνα και είναι και η εφαρμογή αυτής, ε, της, ε, αυτού του σχεδίου δράσης. Ε, μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μα. Έτσι λοιπόν, αν γνωρίζουμε ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και πώ μπορεί να συνεισφέρει η Γεωργία στην επίλυση, πρέπει να αποφασίσουμε ποια Γεωργία θέλουμε για το μέλλον και πρέπει να δούμε ποια Γεωργία μπορεί να, να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτέ τι αλλαγέ. Ε, ε, αυτή η οργία η οποία καταναλώνει νερό, πόρους, υποβαθμίζει το περιβάλλον, καταστρέφει το έδαφος, υποβαθμίζει το τοπίο, τη βιοποικιλότητα και το τοπίο μου θυμίζει αυτό που είπα νωρίτερα ότι ακόμη και αν το τοπίο μπορεί να μην είναι οικονομική αξία, έχει αξία παρόλα αυτά και ποια γεωργία μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το σκοπό. Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα. Μία, ε, ένα παράδειγμα είναι ένα καλά διατηρημένο τοπίο στη Βουργουνδία, όπου έρχεται ένα εξαιρετικό προϊόν που είναι αρκετά ανταγωνιστικό και ταυτόχρονα έχουμε και προστασία του περιβάλλοντος και άλλο παράδειγμα είναι η παραγωγή λαχανικών στη Μεσόγειο με ένα πολύ διαφοροποιημένο περιβάλλον που διατηρεί τις οικολογικές υποδομές ε, και παρέχει και Γη τρόφιμα στους πολίτες. Ε, εδώ αναφέρω τον ορισμό των ε, υπηρεσιών οικοσυστήματος ε, από την έκθεση Millennium και να σας πω ότι δεν παραγεί γεωργία μόνο ε, τρόφιμα, ξύλια κτλ. Αλλά και υπηρεσίε οικοσυστήματο. Και θέλω να υποστηρίξω το εξή. Ενώ έχουμε ένα είδο γεωργία που παρέχει υπηρεσίε οικοσυστήματο, μπορεί επίση ε, να παράσχει και αρκετά ε, ω προ την ποσότητα, δηλαδή τρόφιμα για υγιή τρόπο ζωή. Και εδώ το σχετίζω αυτό μα υποθήκα προηγουμένω από τον πρώτο μιλητή αυτού του πάνελ ότι έχουμε την πρόκληση να πετύχουμε έναν υγιή πληθυσμό στην Ευρώπη και αν θεωρήσουμε ότι η γεωργία μπορεί επίση να συνεισφέρει στην μείωση των δαπανών των κρατών μελών στο να διατηρούνται οι πολίτε υγιεί και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Άλλο σημείο, η Γεωργία μπορεί να συνεισφέρει και στην εξοικονόμηση χρηματών στην περιβαλλοντική προστασία ή στην αναγέννηση του περιβάλλοντος, όπως είπα και πριν. Και κατόπιν αυτού πρέπει να σκεφτούμε, να αποφασίσουμε ποια χειρουργία είναι αυτή που μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτέ τι αλλαγέ, να σκεφτούμε τι γεωργού θέλουμε για να εφαρμόσουν αυτή τη γεωργία. Γιατί μέχρι τώρα συζητάμε την αριστεία στην επιστήμη και πώ θα αξιολογήσουμε την αριστεία στην επιστήμη, πώ θα έχουμε κορυφαία επιστήμη. Αλλά η επιστήμη πρέπει και να εφαρμοστεί μέσω τη καινοτομία ε, και μέσω πράξεων όλων των πολιτών. Έτσι λοιπόν ανησυχώ λίγο περισσότερο για το αν ε, αυτή η επιστήμη αριστεία μπορεί να γίνει ε, στην Ευρώπη καινοτομία αριστεία, η βιολογική, μάλλον όσοι ασχολούνται με τη βιολογική γεωργία μπορούν να εφαρμόσουν ε, αυτή τη γεωργία την οποία αναφέραμε πριν, γιατί είναι νεότερη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με τους συμβατικούς ε, γεωργούς, αυτοί που ασχολούνται με τη βελοκή γεωργία είναι νεότεροι. Μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε στο μέλλον. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι πιο μορφωμένοι, έχουν λάβει καλύτερη κατάρτιση, έχουν ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, μπορούν να εφαρμόσουν λοιπόν καλύτερα την καινοτομία και το αποτέλεσμα τη έρευνα. Ε, είναι εκφύσιος καινοτόμοι γιατί σε ακούσια βάση δέχονται να παράγουν με ένα πιο περιορισμένο και πιο προσεκτικό τρόπο βάσει πρόληψης περισσότερο παραθεραπείας. Έτσι λοιπόν και πάλι ε, τίνουν περισσότερο προς την κοινοτομία και το τελευταίο σημείο είναι ότι απαντούν στο αίτημα των καταναλωτών. Περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ε, το turnover το 2010 για τη βιολογική γεωργία και είχαμε αύξηση στη Γαλλία και στη Γερμανία 10% για τη βιολογική γεωργία. Έτσι λοιπόν μπορεί η βιολογική γεωργία να απαντήσει και στις ανάγκες των πολιτών ε, και στις ανάγκες του περιβάλλοντος, αλλά είναι και ανταγωνιστική από οικονομική σκοπιά. Έτσι λοιπόν αφού αποφασίσαμε ποια γεωργία και ποιους γεωργούς θέλουμε πρέπει να κατανοήσουμε τι καινοτομία και έρευνα χρειάζεται για να υποστηρίξουμε αυτούς τους γεωργούς για να εφαρμόσουν καλύτερα την καινοτομία στα γεωργικά συστήματα και διάλεξα δύο σημεία. Στην ε, ατζέντα μας έχουμε αναπτύξει περισσότερα σημεία, αλλά επέλεξα δύο. Καταρχήν έχουμε την έννοια της οικολειτουργικής αντικοποίησης, δηλαδή να αντικοποιηθεί παραγωγή όχι μόνο τροφίμων, αλλά και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, αλλά με αντίστοιχο τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια καινοτόμο προσέγγιση για να παράξουμε περισσότερο χωρίς ε, να εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους. Έχουμε ήδη λαμπρά παραδείγματα χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για να διευρύνουμε την έννοια και να αντικαταστήσουμε πραγματικότητα σε όλου του τομεί αγροτική παραγωγή. Δεύτερο παράδειγμα, ε, ποικιλότητα από τον αγρό στο πιάτο ή αντιστρόφο. Η ιδέα είναι να ε, χρησιμοποιήσουμε τη βιοπικιλότητα και όλους τους φυσικούς πόρους έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στα τρόφιμα και στα γεωργικά συστήματα. Αν δηλαδή μπορούμε να συνδέσουμε τις δύο προσεγγίσεις μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση κερδοφόρο. Και τι έρευνα χρειαζόμαστε ως προς τη μέθοδο. Τη συμμετοχική μέθοδος ε, τονίστηκε στο παρελθόν. Θέλω να το ξανατονίσω. Χρειαζόμαστε μία προσέγγιση συμμετοχική, αν θέλουμε, επιστήμη της αριστείας να καταστεί πραγματικότητα. Χωρίς αυτό νομίζω ότι χάνουμε μία μεγάλη ευκαιρία. Έτσι λοιπόν, ε, για να προσθέσουμε αυτή την συμμετοχική προσέγγιση και για να μπορεί να εφαρμοστεί παραγωγικά, χρειαζόμαστε ένα δίκτυο τοπικών ε, κέντρων καινοτομία και γνώσης ε, που θα είναι καλά κατανεμημένα σε όλες τις γεωργικές περιοχές. Διαφορετικά δεν θα φτάσουν τα αποτελέσματα στους γεωργού. Και θέλω να τονίσω την ιδέα ότι η γεωργική καινοτομία δεν είναι μόνο ένα νέο προϊόν ή απλά νέα γνώση. Πολύ συχνά αποτελεί συνδυασμό υφιστάμενη γνώσης, παραδοσιακής γνώσης με την καινοτομογνώση είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε για την κοινοτομία στη βιομηχανία, αλλά στη γεωργία ε, έχουμε πολλούς ανθρώπους που την εφαρμόζουμε και ε, διαφορετικά μέσα. Είναι πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν διαφορετικού είδους έρευνας. Αν ήμουν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ θα έθεσα στον εαυτό μου μια ερώτηση. Ποια είναι μια καλή επένδυση των δημοσίων κονδύλιων στην ε, ε, αγροτική έρευνα και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών συστημάτων υψηλής ποιότητα. Δεν υπάρχει ένα σύστημα. Έχουμε πολλά συστήματα που εξυπηρετούν την διαφορετικότητα, την ποικιλότητα της Ευρώπης. Διαφορετικά δεν έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό και ευρωπαϊκή γεωργία, με συγχωρείτε, και ε, αν πρέπει να επενδύσουμε δημόσιου πόρου στην έρευνα για τη γεωργία, θα προσπαθούσα εγώ να δω πώ μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε αυτό το, αυτή την έννοια της εντετικοποίησης, πώς μπορούμε να την καταστήσουμε πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αναφέρθηκε πριν πώς μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία των δράσεων αυτών. Νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε και κάτι σχετικά με την εφαρμογή. Επίσης πρέπει να τονίσουμε τη συμμαχή της ε, κοινωνικής ε, ηγεσίας. Δεν μιλάμε μόνο για τεχνική καινοτομία εδώ, αν έχουμε ένα συνδυασμό υφιστάμενη γνώση με τη νέα γνώση, κοινωνική καινοτομία και οργανωτική καινοτομία μαζί με την τεχνική καινοτομία, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κατάφερα να σεβαστώ το χρόνο, 10 λεπτά και στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα που σας ανέφερα και υπάρχουν και άλλα σχόλια που σχολιάζουν το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Μικελόνη και θα δώσω το λόγο στον Τζον Άντερσεν από το ε, Ίδρυμα της Κοπενχάγης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ε, Πρόεδρο και την Επιτροπή που κάλεσε το Ερευνητικό Κέντρο της Κοπενχάγης για την ε, παρουσίαση αυτή. Το κέντρο μας αναφέρεται σε θέματα συμπληρωματικά που έχουν να κάνουν με την αριστεία που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί. Το κέντρο, το φόρουμ ερευνών της Κοπενχάγης θεωρεί ότι το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 αποτελεί ένα ισχυρό και φιλόδοξο πρόγραμμα για την Ευρώπη. Να σας δώσω μια ιδέα του τι κάνουμε. Το Φόρουμ Ερευνών της Κοπενχάγης αποτελεί μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της ε, Δανίας και συμμετέχουν 600 κορυφαίοι ερευνητές για να, και προσκλήθηκαν για να συνεισφέρουν ως προς πρόγραμμα Ορίζοντες 2020. Να αναφερθώ σε κάτι που αναφέρθηκε στο, σε προηγούμενη φάση. Τρία κριτήρια έπρεπε να πληρούν αυτοί οι 600 ερευνητές. Θα έπρεπε να είναι άριστοι στον τομέα τους από όλη την Ευρώπη και από τα νέα και από τα παλαιά κράτη-μέλη και έπρεπε να υπάρχει και σωστή κατανομή αναφύλο. 16 Ιανουαρίου 2012, 80 ερευνητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στην Κομπεχάγη και κατέκτησαν ε, αυτή τη μελέτη, την οποία και σας ε, μοιράσαμε. Αν μιλάω πολύ γρήγορα, μάλλον θα κοιτάξω σε περίπτωση που δεν καταλάβετε κάτι από τα πορίσματα και τα συμπεράσματα, μπορείτε να τα βρείτε όλα σε έγγραφη μορφή. Οι του λοιπόν του Φόρουμ του Ερευνητικού της Κοπενχάγης παρουσιάστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Φεβρουαρίου του 2012 και αποστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε όλη την Ευρώπη. Ήταν καλή και πολύ ε, θερμή η υποδοχή τους. Ελπίζω και εσείς το ίδιο να θεωρήσετε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα από τα αποτελέσματα, ένα από τα συμπεράσματα του Φόρουμ Ερευνών της Κοπενχάγης είναι ότι ο διατομεακός χαρακτήρας αποτελεί τη βάση της επίλυσης του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Βλέπετε την ε, δημιουργικότητα και τις έντονες συζητήσει που ε, διαμήφθησαν στις 16 Ιανουαρίου. Να περάσω τώρα όπως σας είπα, για κάθε απειλή κοινωνική διοργανώθηκε ένα πάνελ για τον τομέα της υγείας. Ένα από τα πορίσματα ήταν ότι μία από τις βασικές προκλήσεις της Ευρώπης είναι η γύρανση του πληθυσμού με μία σειρά ε, ασθενειών που απειλούν όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και το κόστος που συνεπάγονται για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Μία από τις εξελίξεις που θα διακρίνουμε τα επόμενα 7 χρόνια στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 είναι η εξαρτοφημικευμένη ιατρική. Ένας νέος τρόπος θεώρησης της ιατρικής ε, αναφέρθηκε και προηγουμένως στην εξαιρετική εισήγηση του συναδέλφου. Θα πρέπει να εστιαστούμε εκ νέου στην πρόληψη, στην υγεία εφόρου ζωής και να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματα των μελετών θα μετατραπούν σε καινοτομία για την ανάπτυξη και την υγεία. Στον τομέα της ε, διατροφής των τροφίμων. Κάποιες από τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι ότι χρειαζόμαστε βιώσιμα αποτελέσματα και ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν καινοτομικέ ε, αλυσίδε αξία. Και αυτό είναι συμπληρωματικά προ αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένω, προ τι βασικέ προκλήσει, η σύνδεση μεταξύ τροφίμων και υγεία, διατροφή. Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση της ε, γεωργικής πολιτικής και μία προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη όλο τον κύκλο ζωής θα πρέπει να θεωρούμε ότι τα τρόφιμα και η γεωργία αποτελούν βασικό τομέα για τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρώπη, στον τομέα της ενέργειας. Η μετάβαση σε αξιόπιστα και βιώσιμα και ανταγωνιστικά συστήματα ενέργειας θα πρέπει να κυριαρχεί. Θα πρέπει να οριστεί ένα set plan, θα πρέπει να προσταθεί μια νέα προσέγγιση ε, για έκκληση και ζήτηση για συστημικά και πολυτομιακά προγράμματα ερευνάς θα πρέπει να είναι κατάλληλη χρηματοδότηση στον τομέα των μεταφορών. Βασική πρόκληση, όπως ξέρετε όλοι σας, είναι η πυρεκμετάλλευση των συστημάτων μεταφορών, ε, ε, η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Αυτά είναι τα προβλήματα τα βασικά που μας απασχολούν στον τομέα του κλίματος τώρα. Το πάνελ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα. Θα πρέπει το κλίμα να το θεωρήσουμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάποια από τα βασικά στοιχεία ήταν η χρήση του νερού, ε, η μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, στη βιοπικιλότητα και ούτω καθεξής. Επίσης, στο πάνελ για τις ε, κοινωνικής ε, διαστάσεις υπογραμμίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σωστό, σωστά σημεία βάρους. Αυτό που ήταν πολύ σημαντικό είναι ότι οι κοινωνικές επιστήμες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ατζέντα. Ως εκ τούτου, Υπάρχει μια ξεχωριστή θεωρία που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς όπως ως τώρα, γιατί τώρα τι κάνουμε ουσιαστικά αντιδρούμε σε μια κατάσταση που έχει ήδη διαμορφωθεί. Θα πρέπει στο μέλλον να προγραμματίσουμε εμείς και να διαμορφώσουμε εμείς την μελλοντική κατάσταση. Επίσης, να τονίσω και αυτό που αναφέρθηκε ήδη στο πάνελ, ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να ε, θεωρούνται μόνο ε, καταναλωτές, αλλά και φορείς δράσης. Οι βασικές, λοιπόν, ε, τα βασικά συμπεράσματα του Φόρουμ του Ερευνητικού της Ευρωπαϊκής του είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μία διατομεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Θα πρέπει να συνδυαστεί ο τομέα τη υγεία, τη διατροφή, τη ενέργεια, των μεταφορών, του κλίματο και τη κοινωνική διάσταση και να ενσωματωθούν ο ένας στον άλλον. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση για την μετάβαση σε βιώσιμες κοινωνίες. Εδώ βλέπετε ανεμόμυλους που δεν ε, συμβολίζουν μόνο την ανάγκη για βιώσιμα συστήματα ενέργειας, αλλά παράλληλα υποδεικνύουν ότι όλοι οι μήλοι πρέπει να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα. Τέλος, το φόρουμ της Κοπενχάγης συζήτησε τους ε, όρους πλαίσιο που χρειάζονται. Η αριστεία αποτελεί προϋπόθεση. Επίσης, προκειμένου να δικαιολογηθεί η χρηματοδότηση στα συστήματα έρευνας και ανάπτυξης, χρειάζεται να περάσει η προτινόμενη απλοποίηση του προγράμματος ορίζοντας 2020. Η τελική διατύπωση του προγράμματος θα πρέπει να βρίσκεται με μια, από ένα παγκόσμιο οπτικό σημείο. Χρειάζεται η συμμετοχή όλων των φορέων, των επιχειρήσεων, των ερευνητών, των κρατών και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε πάνω κάτω 20 λεπτά στη διάθεσή μας με τα βίας για τις ερωταπαντήσεις. Θα προτείνω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λαμπέτ, που είναι συνσηγητής για ένα-δυο λεπτά μόνο. Σας παρακαλώ και κατόπιν να ακολουθήσουν οι ερωταπαντήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ στο τελευταίο μιλητή. Συμφωνώ με όσα είπατε για την ε, διατομιακότητα. Έχω μία άμεση ερώτηση για σας. Πιστεύετε ή όχι ότι ο τρόπος που εργάζεται η Επιτροπή, δεν είναι ορθά προσανατολισμένη για να προωθήσει την διατομιακότητα. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς είπατε ότι με τον τρόπο διάρθρωσης ε, των προσκλήσεων, υποβολής προτάσεων, έτσι μπορούμε να φτάσουμε στη διατομιακότητα. Η σημερινή προτινόμενη ε, δομή του προγράμματος ε, και η συνεργασία της Κομισιόν μέσω των διάφορων γενικών διευθύνσεων. Αυτό μας εμποδίζει να φτάσουμε σε αυτή τη διατομεατικότητα. Μήπω πρέπει να υπάρχει εξωτερική ανάθεση των διαγωνισμών σε κάποιον που να εργάζεται ήδη με διατομεακό τρόπο. Ε, οποιαδήποτε σκέψη σε αυτό θα ήταν πρόσδεκτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους ε, ήρθαν να μας μιλήσουν και θα ήθελα συγκεκριμένα να υποβάλω ένα ερώτημα προς τον καθηγητή Σάτοκ από το Imperial. Για πετε μας. Νομίζω ότι το Πανεπιστήμιο σας είχε συμμετάσχει στις ε, συναντήσεις για την αλλαγή του κλίματος και ε, τώρα και εμείς έχουμε προσπαθήσει κάτι να κάνουμε για την, τον τομέα της υγείας. Ε, όντως θέλετε και εσείς χρηματοδότηση, αλλά για να πάρετε χρηματοδότηση θα πρέπει να, ε, να του τους ανταγωνιστές που θέλουν κάτι να γίνει ε, ας πούμε για τις πρώτες ύλες και λοιπά και μιλούμε για ότι, θα πρέπει να βρείτε από κάποιες πηγές 75% και όσον αφορά τις προτεραιότητες αυτές που υπάρχουν ε, και αν πάρτε και το 20% το 70% θα το βρείτε ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν Άλλο θέλει το λόγο λέει ο Πρόεδρος Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την έρευνα, μας αποσχολεί όλους η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. να σας λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονοητό και τελικά αναρωτιόμαστε ως κοινωνία των πολιτών θα τα, θα τα πούμε και με την Επιτροπή το απόγευμα όμως και κοινωνία των πολιτών για μας, δεν έχετε την αίσθηση ότι από κοινού θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε σε κάθε επίπεδο την ε, κρατική χρηματοδότηση, γιατί το έχουμε πει και ξαναπεί, αλλά δεν το λαμβάνω πάντα υπόψη. Θα πρέπει να γίνει μία. Θα πρέπει να γίνει κάποιο και στα τρία επίπεδα. οικονομικός έλεγχο. Περιφέρεια, κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε τι γίνεται με κάποια ποσά τα οποία δαπανούνται και θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερο, καλύτερο, καλύτερο συντονισμός και ίσως θα έπρεπε βέβαια το ελληνικό συνέδριο να κάνει αυτόν τον έλεγχο μαζί με τα 27 εθνικά ελληνικά συνέδρια για να δούμε πώς μπορούμε να αριστοποιήσουμε τους πόρους, τη χρήση των πόρων που έχουμε και σε σχέση με την έρευνα και αν κατάλαβα καλά σε αυτή τη δέσμη προτάσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόταση και το 2012 θα, κάτι θα κάνει όσον αφορά τον ε, ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Άρα θα πρέπει να αναδευτεί κάποια πρωτοβουλία, ε, όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η γενική κατεύθυνση. Τι θέλουμε για το ορίζον 2020 και όλα αυτά τα οποία προτείνονται. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια όσον αφορά επομένω την κρατική ε, παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Ευρώπη, κράτη, περιφέρειες γιατί έχουμε πολλούς πόρους μέσω των, το, μέσο των ιδιωτικών ταμείων. Άρα εσείς τι λέτε, ότι μια που λείπουν τα χρήματα τη σήμερα ημέρα, ε, όσον αφορά τους συμπολίτε μας, προσπαθούμε τώρα να φτιάξουμε αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό για την ανταγωνιστικότητα της Επίρου μας. Ε, Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσε ήταν οι εισηγήσει. Σα ευχαριστώ και να ευχαριστήσω ιδιαίτερω την Βενέζικη Προεδρία γιατί κάλεσε 600 ερευνητέ με μια πρωτοβουλία από όλη την Ευρώπη και έτσι νομίζω ότι έχουμε τους πιο σημαντικούς που από την αρχή να δουλεύουν πάνω σε αυτό. Πολλά χρήματα έχουν ε, διατεθεί προς τούτο γιατί ακριβώς εδώ πέρα δεν θέλουμε διακλαδικότητα, διεπιστημονικότητα και όλα αυτά είναι σημαντικά και για τον τομέα της υγείας και για τη γεωργία είναι σημαντική έρευνα. Για πέστε μας περισσότερα. Τι σχέδια υπάρχουν. Και θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα παράγεται θα παράγονται περισσότερα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερες αγωγές. Το θύμα θα γίνονται η ανιχνευσιμότητα. Ε, σε αυτό είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Και επομένω η έρευνα θα πρέπει να βοηθά, εξασφαλίζει ότι θα έχουμε αυτάρκεια και βιωσιμότητα. Γιατί ό,τι έρχεται από δεν μπορούμε να το ελέγξουμε το ίδιο. Τι θα γίνει επίση και με τη θαλάσσια έρευνα. Πριν από λίγε εβδομάδε έγινε μια έκθεση εδώ και έδειξε τι δυνατότητε που μας παρέχει η θάλασσα. Μας δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία να είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτόν τον τομέα σε σχέση επίσης και με τις διατροφικές ανάγκες. Όλα όσα κάνουμε επομένως στον κλάδο της έρευνα θα ωφελήσει, σε δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Επομένως, διαπέστε για τη γνώμη πάνω σε αυτά. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Επομένω, στα επόμενα δέκα λεπτά που μα μένουν, να επιτρέψουμε στου ομιλητέ να απαντήσουν και να δώσουμε και δύο λεπτά στην συνάδελφο για τα συμπεράσματα. Λοιπόν, ο κύριο Σάτοκ, ο καθηγητή Σάτοκ και θα σα δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θέλω να απαντήσω καταρχήν στην ερώτηση για το αν ένα παρόμοιο μοντέλο με αυτό που εφαρμόζεται στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ορισμένες ανάγκες ε, στον τομέα τη υγεία και ιδίω για τι ενώσει που σχετίζονται με τη φτώχεια. Νομίζω ότι είναι καλό μοντέλο. Τώρα θα έχουμε μια σημαντική πρόκληση να συγκεντρώσουμε το 75% της χρηματοδότησης, μπορεί να μπορέσουμε ε, να συγκεντρώσουμε το 50% από μια καινή πρόταση χρηματοδότησης. Αυτό σίγουρα θα είναι κάτι δυνατό και ελκυστικό και νομίζω ότι αυτό τονίζει και την κατακαιρματισμένη φύση της έρευνας ε, στις ε, νόσους που σχετίζονται με την φτώχεια, με την ενέχεια σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ε, και στα ευρωπαϊκά αλλά και στα εθνικά προγράμματα και πολλές φορές σε διεθνές επίπεδο βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει μια ισχυρή φωνή σε ό,τι αφορά αυτές τις νόσους ε, που σχετίζονται με την ανέχεια. Ε, δεν υπάρχουν πάρα πολλέ ομάδε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που να ασχολούνται με αυτέ τι νόσου. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να προσδώσουμε προσοχή σε αυτό το τομέα για το πώ θα προωθήσουμε την ευρωπαϊκή αριστεία σε διεθνέ επίπεδο σε ό,τι αφορά την έρευνα στον τομέα της υγείας και θέλω να κλείσω απλώ τονίζοντας τη συνεχή ανάγκη για κατάρτιση στον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε νέα γενιά ερευνητών που να μπορούν να εργαστούν ε, τομέα αυτών των νόσων που σχετίζονται με την ανέχεια, αλλά δεν αρκεί να επενδύουμε ε, σε ε, κάποια συστήματα μεταδιδακτορικά μόνο, γιατί δεν παρέχεται ασφαλεία σταδιοδρομίας έτσι στους ερευνητές. Πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, για να μην δημιουργούμε λοιπόν απλώ συστήματα κατάρτιση όπου κάποιοι επενδύουν 10-15 χρόνια τη ζωή του, αλλά κατόπιν πρέπει να εγκαταλείψουν την επιστήμη γιατί δεν υπάρχουν βιώσιμε προοπτικέ πέραν αυτού. Η κυρία Κλάουδια Νόιμπερ. Mm-hmm. I would maybe, um, starting from... Θα ξεκινήσω από την γαλλική ερώτηση, να το θέσω έτσι. σας προτείνω κάποιες σκέψεις για την καινοτομία. Δηλαδή, ποια ερμηνεία και ποια κατανόηση έχουμε σήμερα όταν ακούμε τον όρο καινοτομία. Ας πούμε ότι σήμερα έχουμε την τάση όταν ακούμε καινοτομία να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για ε, υψηλές τεχνολογικές εξελίξεις ή για υψηλά τεχνολογικά προϊόντα και όχι τόσο ε, για προϊόντα που δεν σχετίζονται με τεχνολογία. Πρόκειται για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία και ίσω να δώσουμε λιγότερο χώρο στην ε, ανοιχτή πρόσβαση στα αποτελέσματα. Επίση, ε, είναι θέμα της ε, προσβασιμότητας σε τι πρόσβαση έχουν σε αυτή την καινοτομία περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί. Έχει να κάνει με το επίπεδο παρέμβαση της καινοτομία περισσότερο σε παγκόσμιο ή τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, να πρέπει να σκεφτόμαστε σε τοπικό επίπεδο και να αποκεντρώνουμε την αγιοργία, την ενεργειακό φεδιασμό κτλ. Επίσης, ε, για τον ορίζοντα 2020 πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό με υψηλό επίπεδο έρευνα και καινοτομία. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε υψηλό επίπεδο κινδύνου, ανάληψη ε, κινδύνου στην καινοτομία και φυσικά αυτό προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αν σκεφτούμε τι έγινε με μια τελευταία δημοσίευση ερευνητών που εργάζονταν για ένα θέμα που ε, ήταν ε, πάρα πολύ επικίνδυνο και μπλοκαρίστηκε η δημοσίευσή τους. Και μιλάμε για πάρα πολύ ταλαντούχους ερευνητές, αλλά μια τέτοια έρευνα τι να τη κάνουμε. Επίσης, ε, είπα ότι δίνουμε στην κοινωνία των πολιτών ε, και στη βιομηχανία ε, τι ρόλο προσδίδουμε και υπάρχει μεγάλη ανισορροπία σήμερα. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη επικέντρωση στις ΣΔΙΤ και όχι στους άλλους πρωταγωνιστές πέραν της βιομηχανίας. Και επίσης, δεν έχουμε συζητήσει αρκετά το θέμα του προσωρίζουμε την επιστημονική αριστεία τουλάχιστον στην Γαλλία σήμερα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων, με ποια κριτήρια πρέπει να καθορίσουμε την επιστημονική αριστεία. Όπως ξέρουμε σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο σε ορισμένους επιστημονικούς τομείς να πάρει κάποιο βρεβείο για επιστημονική αριστεία παρά σε άλλους και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μικελώνη. Thanks. ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω τρία ζητήματα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το τέλος, για θέματα υγείας και σύνδεσης μεταξύ διατροφής, παραγωγής τροφίμων και γεωργίας και το θέμα της πιο έντονης ευρωπαϊκής παραγωγής ε, τροφίμων και ζωοτροφών, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές ε. Είναι καλέ οι προοπτικέ για την ανάκτηση τομέων που είχαν περιθωριοποιηθεί προκειμένου να συμβάλλουν στην καλύτερη παραγωγή για τρόφιμα και ζωοτροφές για να καλύψουν τις τοπικές αγορές αλλά και για την αναζωγόνηση των κοινοτήτων. Το δεύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας και σε ό,τι αφορά τη βιολογική παραγωγή, για παράδειγμα, γίνονται προσπάθειες να συγκεντρωθεί η γνώση και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες. Θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο μεγάλης βελτίωσης, αλλά πρόκειται για μια ανησυχία η οποία έχει ήδη εντοπιστεί και αντιμετωπίζεται και νομίζω σημαντικό θα είναι πώς θα δημορφωθεί και η καινούργια ΚΑΠ από το 2013, γιατί εκεί για τη γεωργία σε κάθε περίπτωση αίτησης αρρωγής θα πρέπει να ε, καταδειχθεί το τεχνικό επίπεδο της ε, αίτησης. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν να συνδυάσουμε το πρόγραμμα Ορίζοντες 2020 με την ε, νέα ΚΑΠ, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η δαπάνη πολλών πόρων. Ίσως πιο πολλές ε, ε, αιτήσει στα πλαίσια της Aranet. Για το τελευταίο ζήτημα, της διατομεακότητας. Ε, δεν το ανέφερα στην εισήγησή μου, αλλά βασικό είναι να υπάρχει εφαρμογή σε δύο τομείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ πρόβλημα στις αιτήσει, αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στην ευρωπαϊκή πολιτική, ότι δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή με διατομιακό τρόπο όλα αυτά. Ε, ε. ευχαριστούμε και ο κύριος Άντερσεν για την τελευταία παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσω κι εγώ από εκεί που τελειώσατε. Πώς Νομίζω ότι χωρίς να είμαι εμπειρογνώμων, πρέπει να πω ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να παράγει τα τρόφιμα που χρειάζεται το πληθυσμό της. Αλλά θα ξέρετε ασφαλώς ότι υπάρχει ένα όριο σε ό,τι αφορά την απόδοση, ένα εμπόδιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια σωστή και εντελεχής μελέτη για το πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό το εμπόδιο απόδοσης, προκειμένου όμως να παραμείνει η βιώσιμη παραγωγή. Γιατί υπάρχουν και περιορισμοί σε ό,τι αφορά την υγεία, τη χρήση του νερού και το καθεξής. Ήταν συνάδελφος. Αυτό περιλαμβάνει και την θαλάσσια έρευνα. Με ρωτήσατε επίσης αν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να επιλύσει μάλλον να εφαρμόσει μια διατομιακή προσέγγιση. Πριν από ένα χρόνο, με είχατε ρωτήσει, θα ήμουν πάρα πολύ διδακτικό στην απάντησή μου. Αλλά αυτό που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα Horizon 2020 κατά τίτραση στις συστάσεις που τους ε, δόθηκαν, θεωρώ ότι αποτελούν μια πραγματική δέσμευση για πραγματική προσπάθεια εφαρμογής, εφαρμογής του διατομιακού χαρακτήρα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτός ο διατομεακός χαρακτήρας θα πρέπει να οριστεί καλύτερα. Υπάρχουν πολλοί τύποι διατομεακού χαρακτήρα και υπάρχουν και κάποια πρακτικά εμπόδια, γιατί συχνά τα πάνελ αναθεώρησης ε, περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς τομείς, άρα παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως τα project. Η βασική μου όμως ανησυχία δεν έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εξωτερικής φύσεως, γιατί αυτά που βλέπουμε εξωτερικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι υπηρεσίες δημιουργούν νέους κανόνες και κανονισμούς και μας προκαλούν εφιάλτες σε ό,τι αφορά την υποστήριξη και την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή πρέπει να πω ότι έχω πίστη στο ότι θα μας ακούσει και θα μας εισακούσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα βρει νέους τρόπους επίλυσης των ζητημάτων. Προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη βοηθήσουμε για την κατάρτιση νέων μοντέλων μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και για την τελική σας πρόταση. Λοιπόν, τώρα το λόγο στην κυρία Ματίας για τα συμπεράσματα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Και θα ήθελα να πω ότι είχαμε δύο πολύ διαφορετικά πάνελ ε, για την αριστεία και για την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι θέλουμε, ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε πιο εγγύης αυτές τις δύο έννοιες. Ε, η κυρία Ματίας, ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά κατά εξαίρεξη, προκειμένου να είμαι το συντομότερο δυνατή, το δυνατόν συντομότερη να ευχαριστήσω όλους τους καλασμένους μας για τη συμμετοχή τους και θα ήθελα να τονίσω βασικά τα δύσκολα ερωτήματα τα οποία έθεσαν και έθεσαν επιτάπητος τις εισηγήσεις τους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες άλλωστε. Θα έχουμε χρόνο να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι τέσσερις παρουσιάσεις μας ε, μετέφεραν βασικά τέσσερα μηνύματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε στη διάρκεια επεξεργασία του προγράμματος Horizon 2020. Το πρώτο είναι το θέμα της υγείας, η πρόκληση της υγείας, οι καθολικέ προκλήσει της υγείας. Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε, να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ότι υπάρχουν παγκόσμιες προκλήσεις στην υγεία Θα πρέπει να δώσουμε νέες εμφάσεις στο έργο μας για να ανταποκριθούμε στα νέα αναδυόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε από το μηδέν σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέχεια, κάποια ε, διαρκής βάση, προκειμένου να προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στις νέες προκλήσεις που αναδύονται υπό του νέους όρους που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα παλιά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, τα νέα αναδυόμενα προβλήματα και νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά με τα παραδείγματα του HIV και της θυματίωσης. Να σας ευχαριστήσω που το θέσατε, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να τα αγνοούμε να εξετάζουμε νέες προκλήσεις παραμελώντας τι παλιέ. Είναι τεράστια σημασία λοιπόν αυτή η συνέχεια. Το δεύτερο βασικό και δύσκολο ζήτημα είναι αυτό που έθεσε η Κλάουντα Νόιμπαουερ και έχει να κάνει με το ότι το πρόβλημα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρόγραμμα Horizon 2020 θέτει ένα παράδειγμα το οποίο είναι ήταν σημαντικό στη δεκαετία του 90, αλλά δεν είναι πλέον τόσο σημαντικό. Το παράδειγμα της ε, δημόσιας κατανόησης ε, της ε, επιστήμης από το κοινό. Λέγαμε ότι το κοινό δεν μπορεί να συνεισφέρει τίποτα στην επιστήμη και στην έρευνα, μόνο να λάβει Μετά όμως ε, διαμορφώθηκε η ιδέα της δημόσιας συμμετοχής της επιστήμης. Αν λοιπόν αντιμετωπίζουμε κοινωνικές ε, προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κοινωνίας και των πολιτών και αυτού που συμμετέχουν, αυτών προς τους οποίους θέλουμε να στραφούμε για την επίλυση των προβλημάτων τους. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί το βασικό μας στόχο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των κοινωνιών, των πολιτών. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν την πτυχή των πολιτών, την πτυχή της κοινωνίας. Τρίτο ζήτημα, το οποίο έθεσε η Κριστίνα Μικελάνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο. Το ανέφερε σε ό,τι αφορά την Γεωργία. Μας ρώτησε τι είναι καλή επένδυση όταν μιλάμε για τη γεωργία. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα εγκάρσιο ε, ζήτημα, εγκάρσιο ερώτημα. Τι αποτελεί καλή, καλή επένδυση όταν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Θα πρέπει να το απαντήσουμε το ερώτημα αυτό, γιατί αυτό είναι που μας απασχολεί στην τελική ανάλυση. Τέλος και σε σχέση με αυτά τα ζητήματα τα δύσκολα, νομίζω αυτό το θέμα που έθεσε ο Γιάνν Άντερσεν έχει να κάνει με αυτά είναι το εξή θέμα. Μιλώντας για δημόσιες επενδύσεις και διατομιακό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το πλέγμα των τεράστιων ε, κοινωνικών προκλήσεων, δεν μπορούμε να μπλέξουμε την ε, απλοποίηση με την μείωση, αν θέλετε, του περίπλοκου χαρακτήρα της κοινωνίας. Γιατί αυτό θα αποτελούσε μια παγίδα στην οποία δεν θέλουμε να πέσουμε. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι για τις παρεμβάσεις σας. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας αναφορικά με τις προκλήσεις που μας αναφέρατε και λυπάμαι που ήμουν τόσο σύντομη σε ό,τι αφορά την ανακεφαλαίωση των πολύ σημαντικών αυτών στοιχείων που μας παρουσιάσατε. Ελπίζω να συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές και σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ όλους και εγώ. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες και τους συνοδέλφους και φυσικά όπως ξέρετε θα τα ξαναπούμε στις 3.